So, herzlich willkommen zu unserer... Καλώς ήρθατε, λοιπόν θερμά στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής μας για φέτος. Στην ημερήσια διάταξη έχουμε μια μικρή αλλαγή, το σημείο 11, θα με το 10, μικρή αλλαγή. Έχει να κάνει με τη διαθεσιμότητα των ε, συντακτών. Σημείο 2 Έχουμε όλες τις γλώσσες εκτός από μαλτέζικα, κροατικά και γοεδελικά. Στη συνέχεια έχετε μια σειρά ενημερωτικά σημειώματα για τις αντιπροσωπείες των περασμένων εβδομάδων. Στις κάτω χώρες ήταν η πρώτη αποστολή που ασχολήθηκε με την επερχόμενη Προεδρία για την ίση αμοιβή για ίδια εργασία στον ίδιο χώρο εργασίας. Το πακέτο κινητικότητα, επίσης που θέλει να προωθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αλλάξει η κατάσταση στο μεταξύ και αυτή την εβδομάδα θα υπάρξει και μια μικρή συζήτηση Μήπω αλλάξουν οι προτεραιότητες της ε, Ολλανδική Προεδρία. Προεδρίας. Μετά, καταπολέμηση της ένδυα και του κοινωνικού αποκλεισμού επίσης μας απασχόλησε το θέμα της ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία, ιδιαίτερα για τις καρκινογόνες ουσίες κτλ. Δεν χρειάζεται τώρα να μπαίνω σε λεπτομέρειες, τα έχετε στα χέρια σας στο ενημερωτικό σημείωμα. Την ίδια εβδομάδα ε, μετέβει αποστολή στη Γενέβη στο Διεθνή Οργανισμό Εργασίας. Είναι μια πάγια και καλή ε, παράδοση πλέον της Επιτροπής μας. Ε, ημερήσια αποστολή με πολύ εντατικές επαφές, ιδιαίτερα για το πώς θα ενταχθούν οι πρόσφυγες στην αγορά εργασίας, τι κάνει το γραφείο αυτό, ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας στην Ελλάδα. Συζητήσαμε την ψηφιοποίηση και το μέλλον της εργασίας, ενδιαφέρουσα ενημέρωση. Στο επόμενο ετήσιο συνέδριό τους θα προετοιμάσουν έτσι, κάτι ένα ψήφισμα για το θέμα των ε, ε, αλυσίδων ε, παραγωγής και προσφοράς και θέματα δεοντολογίας. Την ίδια εβδομάδα την προσωπία στην Πορτογαλία ορισμένα μέλη της Επιτροπής μας που συζήτησαν την κατάσταση εκεί, ιδιαίτερα τα θέματα τα κοινωνικά και της απασχόλησης, σε μια χώρα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος προσαρμογής την περασμένη εβδομάδα επίσης είχαμε μία αποστολή ε, για την Ελλάδα που είχαμε αποφασίσει για παρακολούθηση. Αλλά παρακαλώ να το συζητήσουν αυτό οι συντονιστές ε, για πρώτη φορά σήμερα. Τελευταία παρατήρηση στις ανακοινώσεις θα ήθελα να σας πω ότι το βράδυ μετά τη συνεδρία των συντονιστών μας εδώ στον τρίτο όροφο θα έχουμε ε, την ετήσια δεξίωσή μας αποχαιριστική χριστουγεννιάτικη στο όλοι προσκεκλημένη θερμότατα. Πάμε λοιπόν στο σημείο τώρα του προϋπολογισμού. Εκεί έχουμε συνοψίσει όλα τα θέματα όχα, ε, γεροφάν και τεντεφόπ Ο David Κάζα που είναι αρμόδιος συντάκτης ε, κολλείεται και θα τον εκπροσωπήσει ο Ζόρς Μπαχ για πέντε λεπτά, μέσα σε πέντε λεπτά αν γίνεται, να τα χωρέσεις. Σήμερα μιλώ αγγλικά εξ ονόματος του κυρίου Κάζα. Ο οποίος δεν μπορούσε να έρθει στη συνεδρίαση. Θα δοκιμάσω στα αγγλικά. Ο κύριος Κάζα έχει ετοιμάσει και ένα σχετικό σημείο μας στα αγγλικά θα σας το παρουσιάσω. Η Επιτροπή μας θα συντάξει έξι νομοδοτήσεις για τις απαλλαγές του 2014, για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ιματρία, για τους εκτελεστικούς οργανισμούς και τις ε, διοικητικές διαδικασίες, για τους οργανισμούς που έχουν να κάνουν με την απασχόληση. Όπως είπατε, το ETF, το SEDEFOP, το Eurofound και το NOSA. Επίσης θα δούμε τις επιδόσεις, την οικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των ευρωπαϊκών οργανισμών. Τα έγγραφα θα είναι περίπου μια σελίδα στο καθένα και μερικές παρατηρήσεις από τις θυμοδοτήσεις που θα πρέπει να μας απασχόλησουν. Πρώτα απ' όλα η απαλλαγή για την εκτέλεση του Γενικού Προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το δημοσιονομικό έτος 2014 η γνωμοδότηση αυτή σε γενικές γραμμές αντικατοπτρίζει τα πορίσματα των κεφαλαίων 5 και 6 της ετήσιας έκθεσης του ελληνικτικού συνεδρίου για την εκτέλεση του προπολογισμού για το δημοσιονομικό έτος 2014 μαζί με τις απαντήσεις των θεσμικών οργάνων. Κάποιες παρατυπίες έχουν ε, εντοπιστεί από τις μικρομεσαίες την προετοιμασία του προγράμματος Ορίζοντα 2020, αλλά αυτά καλύφθηκαν από την απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό το καλωσορίζουμε δεδομένες της οπτικής σημασίας της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πρόγραμμα για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξης. Η σημασία της καλύτερης χρήσης της ε, απλούστευσης της διαδικασίας για τις νομοτήσεις ε, σημειώνεται και για να μειωθεί το διοικητικό άκθος για τους δικαιούχους. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακολουθήσει τις πρόσφατες συστάσεις του συνεδρίου, του ελεγκτικού συνεδρίου, για να βεβαιωθεί ότι η εκτέλεση του ευρωπαϊκού προπολογισμού συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής του 2020 για την απασχόληση για τις τέσσερις εργασίες. Κάποια στοιχεία της εκτέλεσης τώρα για τους τέσσερις οργανισμούς. Πρώτα απ' όλα το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής ε, Εκπαίδευσης. Η δημοσιονομική του θέση είναι πολύ σημαντική και οι επιδέσεις του επηρεάζονται ε, σχετικά κατά 97% στους τρεις στρατηγικούς στόχους που συνδέονται με την επαγγελματική εκπαίδευση και τα θέματα κατάρτισης. Έχουμε σημειώσει ότι το επίπεδο ε, ανάληψης υποχρέωσεων είναι υψηλό, αλλά αυτό μπορεί να βελτιωθεί με καλύτερες οικονομικές προβλέψεις στο, δημοσιονομικές προβλέψεις στο μέλλον. Επίσης ένα σχετικό βαθμός ευελιξίας χρειάζεται λόγω της δυναμικής εξέλιξης του περιβάλλοντος εδώ στο οποίο λειτουργεί το ETF, ιδίως για το 2014 όπως ήταν τα πράγματα και λόγω της πολιτικής αστάθειας στις χώρες που συμμετέχουν στην πολιτική γειτονία. Για το ΣΕΝΤΕΦΟΠ ε, η αποτίμηση εδώ είναι θετική και η γνωμοδότηση λόγω της κεντρικής ε, οικονομικής θέσης και τον υψηλό βαθμό εκτέλεσης του προπολογισμού. Ε, απορρόφησης δηλαδή. Είναι σημαντικό να σημειώνουμε ότι επικεντρώνεται στο να στηρίζει συμπληρωματικέ πολιτικές για την ανεργία των νέων λόγου χάρη, καθώς και τις δεξιότητες για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Επίσης υπογραμμίζεται στην νομοδότηση ότι υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις για τις επισκευές του κτηρίου του κέντρου που δεν επιτρέπουν ε, ε, δεν επιτρέπει αυτή η καθυστέρηση να αξιοποιήσει πλήρω τι δυνατότητέ του το κέντρο ακόμη. Επίση, είναι γενικώ θετική η αποτίμηση για το ίδρυμα, το Eurofound, που παραμένει ένα από του βασικού συμβάλλοντε στην πολιτική, στη χάραξη πολιτική και την αξιοποίηση τη εμπειρογνωμοσύνη που διαθέτει στα βασικά έγγραφα τη Ευρωπαϊκή Ένωση οι βασικοί δείκτες επιδόσεων όπως η υψηλή ορατότητα και η προβολή των ερευνών είναι σημαντικά στοιχεία. Επίσης καλωσορίζουμε το γεγονός ότι το Eurofound συνεχίζει να επικεντρώνει τις ερευνές του στην αντιμετώπιση της ενεργείας των νέων. Και καλωσορίζουμε τις διχοτικές δράσεις λόγω των μεριμνών που εντέπισε, εντόπισε το ελεγκτικό συνέδριο σε σχέση με τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και την καταγραφή τους. Πρέπει να υπάρξει μια σωστή συμφωνία μεταξύ του Eurofound και της χώρας που υποφιλοξενεί για να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια στις διαδικασίες αυτές. Για τον ΩΣΑ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, και εδώ είναι θετική αποτίμηση, η το ποσοστό απορρόφησης και εκτέλεσης του προπολογισμού ήταν καλό και επίσης ήταν και το πρώτο έτος του πολιετού στρατηγικού προγράμματος του οργανισμού για τα έτη 2014-2020. Είναι θετικές οι ενδείξεις για τα επιτεύγματα του οργανισμού στο πρώτο αυτό έτος, στις ε, τομείς προτεραιότητας όπως ορίζονται στη στρατηγική. Και καλωσορίζουμε στο θετικό βήμα την ανακαίνιση των εγκαταστάσεων και τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί με τις Ισπανικές Αρχές. Η απαλλαγή για την εκτέλεση του προπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2014, καθώς και οι επιδόσεις, ο, η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος των οργανισμών, η γνωμοδότηση αυτή αναφέρεται στους ε, τρεις οδικούς χάρτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουν να κάνουν με την αναθεώρηση των κανονισμών των ε, τριμερών αυτών οργανισμών της Ευρωπαϊκής είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί ο τρομερής χαρακτήρα των οργανισμών και οι σχέσεις συνεργασία, ο συντονισμό και η αμοιβαιότητα στην εργασία των, ε, η συμπληρωματικότητα των οργανισμών πρέπει να διαφυλαχθούν. Θα ήθελα να τονίσω ότι η προθεσμία για την υποβολή των είναι 14 Δεκεμβρίου 2015. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Ζώσο πάντα ευσύνοπτα και σαφή αυτά που μας λες. Ευχαριστώ πολύ. Ο Γκριγόρ Γιώργη Πυρίνσκη, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Uh, ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πάρα πολύ τον εισηγητή κατάργο του. Οι προτάσεις του είναι σωστές, όπως συμπεριλαμβάνονται στις διάφορες απαλλαγές για την Επιτροπή αλλά και για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς. Όσον αφορά την απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πράγματι είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι η απλοποίηση έχει μεγάλη σημασία και κυρίως όσον αφορά το κόστος. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του ελεκτικού συνεδρίου, είναι προτιμότερη απλοποίηση και θα έπρεπε να θαρρυνθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το κάνει. Θα πρέπει στις διαχειριστικές αρχές να δίνει τις κατάλληλες κατευθυντήριες γραμμές για να μπορούν να επιλέγουν σωστά και για το διάστημα 2014 με 2020 μπορεί έτσι να γίνει εξοικονόμηση. Οι χώρες μέλη σε εθνικό επίπεδο δεν πρέπει να περιπλέκουν τα πράγματα όσον αφορά την χρήση των κονδυλίων του κοινωνικού ταμείου. Γιατί τότε οι δικαιούχοι επιβαρύνονται επιπλέον και υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος φάλματος. Προτείνω επίση να θαρρύνουμε τις χώρες μέλη να χρησιμοποιούν το εργαλείο Εράκνη όσον αφορά την αξιολόγηση κινδύνου και να δίνουν τις σωστές κατευθυντήριες γραμμές στις χώρες μέλη και την τεχνική αρρωγή για την εφαρμογή των απαιτήσεων όσον αφορά τη διαχείριση και τον έλεγχο για την περίοδο 2014-2020. Πρόκειται για θέμα καλών πρακτικών μεταξύ των χωρών μελών. Τώρα στην ετήσια εκθέση του ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρεται ότι Υπάρχει αύξηση των δικτών όσον αφορά τα κοινωνικά ζητήματα σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Και στι παρατηρήσει του Ελληνικού Συνέδριου λέει ότι το ποσοστό σφάλματος θα ήταν χαμηλότερο αν οι εθνικέ αρχέ είχαν χρησιμοποιήσει τι πληροφορίε που υπάρχουν πριν στείλουν στην Επιτροπή αιτήσει για πληρωμέ. Συνεπώς, οι χώρε μέλη πρέπει να ελέγχουν καλύτερα τα πράγματα και να μην ζητούν αποζημιώσει για ε, πληρωμές που κανονικά δεν πρέπει να γίνουν. Επίση, άλλη σύσταση του Ελεκτικού συνεδρίου είναι οι χωρε μέλη να πληρώνουν τους δικαιούχου πιο γρήγορα, σύμφωνα με τα χρονοδιάγραμματα που προβλέπονται στου κανονισμούς. Τώρα, για τα αποτελέσματα και την επίτευξη των στόχων στις κοινωνικές επιθέσεις για την περίοδο 2014-2020 ελπίζουμε να υπάρχουν καλύτερες επιδόσεις και κυρίως καλύτερη αναφορά των επιτευγμάτων που θα έχουμε την περίοδο αυτή. Τώρα πιο συγκεκριμένα για τα ιδρύματα και τους οργανισμούς. Γενικά όσον αφορά τις επιδόσεις τους, την διαχείριση και τον έλεγχο για το 2014, στηρίζω την εφαρμογή του χάρτη πορείας και των δράσεων που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2014 δεν έχουν ε, ολοκληρώσει τις δράσεις τους όλοι οι οργανισμοί και τα ιδρύματα, γι' αυτό προτείνω να πιέσουμε τους οργανισμούς που δεν έχουν ακόμα τα κατάλληλα πλαίσια με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να το πράξουν. Να επιμείνουν επίσης να προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους εφόσον δεν έχουν ε, στρατηγική κατά των απατών και αυτό να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και όσον αφορά τους δείκτες επιδόσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να τους εφαρμόσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα και οι κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την εφαρμογή των ε, κανόνων να ακολουθήσουν την αρχή της απλοποίησης για να εξοικονομήσουμε χρόνο και χρήμα. Καλώς ορίζω επίσης και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών. Λαμβάνουμε υπόψη μας και τα σχόλια του ελεκτικού συνεδρίου όσον αφορά την χρήση προϋπολογισμού από τους οργανισμούς όσον αφορά τα carry overs των ε, υποχρεώσεων συχνά τα αποτελέσματα αυτά ε, σημαίνει ότι ε, ξεφεύγει ο έλεγχος μερικές φορές από τους οργανισμούς. Δικαιολογείται μερικές φορές επειδή διάφορες δραστηριότητες είναι πολυετής οι προγράμματα. Όσον αφορά τώρα τις ε, διάφορες γνωμοδοτήσεις, προτείνω να σχολιάσουμε τα αποτελέσματα για το 2014 συμπεριλαμβάνοντας τις επιπτώσεις στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά το Ίδρυμα επαγγελματική Εκπαίδευσης, προτείνω συντονισμό των δραστηριοτήτων στις διάφορες χώρες με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και για το κέντρο για την ανάπτυξη επαγγελματικής κατάρτισης, εδώ υπάρχει και το θέμα των ε, προσφύγων που θα επηρεάσει τις δραστηριότητες και το σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια. Θα προτείνω διάφορες τροπολογίες και προσβλέπω σε συνεργασία με τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές για την απαλλαγή 2014. Ευχαριστώ. Από τους συντηρητικούς ε, και μεταρρυθμιστές κανονικά ο κύριος Μπασίρ, αλλά μάλλον τον εκπροσωπεί άλλος συνάδελφος. Ευχαριστώ εκ μέρου του κυρίου Μπασίτ. Να πω ότι με ικανοποίηση σημειώνω ότι το ποσοστό εκτέλεση, το ποσοστό μάλλον αρνητικών σχολείων έχει χαμηλώσει πολύ, αλλά ακόμη δεν είναι αρκετό. Το ποσοστό σφάλματο έχει αυξηθεί στον τομέα τη απασχόληση και των κοινωνικών υποθέσεων. Ε, η έκκληση του κυρίου Κάζα για αυστηρότερε διαδικασίε για να μειωθεί ο κίνδυνο παρατυπιών σε αυτό το τομέα πολιτικής είναι πολύ εύστοχη. Η ομάδα μου αναμένει την έκθεση για την πρωτοβουλία για τους νέους της Ευρώπης και το Ταμείο Γύσης για τους νέους διότι θεωρούμε ότι ακόμη δεν έχει γίνει επαρκής χρήση των ε, διατηθέμενων κονδύλιων. Επίση, οι στόχοι που προβλέπονται από τα κονδύλια τη Ένωση για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, είναι πολύ σημαντικέ για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτέ τι κινητήριε ε, μηχανέ για την ανάπτυξη που πρέπει να υποφεληθούν από τα κονδύλια όπω και μεγαλύτερε εταιρείε. Είναι σημαντικό πάντω να ενθαρρύνουμε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει να συμμετέχουν σε προγράμματα χρηματοδότηση, όπω το Horizon 2020 και το ERDF ε, με μικρότερα ποσοστά σφάλματος. Πρέπει να βρεθεί το κατάλληλο σημείο ισορροπίας εδώ για να είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρχει κατάλληλο σύστημα για τη μείωση των προτυπιών και ότι αυτό θα ισχύσει χωρίς να παρεμποδιστεί η μεγαλύτερη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι συντηρητικοί και μεταρρυθμιστές καλωσορίζουν τις κινήσεις για την βελτίωση της πολιτικής και ανάλογε κινήσει προ αυτή την κατεύθυνση. Ω προς τους οργανισμούς θεωρούμε ε, ανέκαθεν ότι ο μεγάλος αριθμός ε, οργανισμών που υπάρχουν δεν είναι απαραίτητο και υπάρχει επικάλυψη στις εργασίες πολλών από του οργανισμού. Ένα παράδειγμα για αυτά είναι το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και το Ευρωπαϊκό ε, Ίδρυμα για την Κατάρτιση για την ανάπτυξη της επαγγελματική κατάρτισης, ο DEFOP και η ETF. Θα μπορούσαν να συγχωνευτούν αυτές οι δύο περιπτώσεις, αυτά τα δύο οργανισμοί, ώστε να έχουμε και καλές εξοικονομήσεις. Ευχαριστώ τον κύριο Κάζα και θα φροντίσουμε ως συντηρητικοί μεταρρυθμιστές να υποβάλουμε κάποιες τοπολογίες για τα ζητήματα που έθιξε. Ευχαριστώ πολύ. Και εκ μέρους του κυρίου, του κυρίου φυσικά. Ευχαριστώ πολύ. Από του η Μάριαν Χάρκινγκ η επίσης και απουσιάζει. Κανονικά η κυρία Μπόιλαν, την οποία και δεν βλέπω, και κανέναν άλλον ε, άλλος από άλλη πολιτική ομάδα, η FTT, κανένα, η ΕΝΕΦ, Ντομινίκ Μαρτά απουσιάζει επίσης, ε, απίστευτη με διαδικασίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Thank you very much for the, for the floor, Mr. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα σας μιλήσω για το γενικό θέμα της απαλλαγής και αν χρειάζεται ο συνάδελφος θα συμπληρώσει για τους οργανισμούς και τα ιδρύματα. Εγώ είμαι από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και είμαι υπεύθυνο του τμήματο Απαλλαγής. Χαίρομαι για το σχέδιο αυτό έκθεσης του εισηγητή που τονίζει και υπογραμμίζει τα διάφορα ζητήματα που και εμείς βλέπουμε στη... στο θέμα αυτό της απαλλαγής και θέλω να σχολιάσω δύο ζητήματα τα οποία αναφέρονται στις γνωμοδοτήσεις. Πρώτον, υπογραμμίζω τη σημασία που δίνουμε και εμείς σε παρετέρω απλοποίηση, κυρίως όσον αφορά την ενίσχυση της χρήσης των επιλογών ε, απλοποιημένου κόστους. Όπως πολύ σωστά είπε και ο κύριος Πυρίνσκι και αναφέρεται και υπογραμμίζεται και στην γνωμοδότηση αυτή. Ενώ λοιπόν είναι αλήθεια ότι οι απλοποιημένες αυτές ε, διαδικασίες ελαφρύνουν το διοικητικό άχθος, συγχρόνως κατά τη γνώμη μας συνεισφέρουν στη μείωση του ποσοστού σφάλματος. Και κυρίως και πιο σημαντικό ακόμα μας επιτρέπουν να επικεντρωνόμαστε περισσότερο στα αποτελέσματα και στις επιδόσεις. Γιατί οδηγούν σε αποζημιώσεις που έχουν να κάνουν με τα αποτελέσματα που έχουν επιτεθεί. Δεύτερον, επίσης αναφέρεται στη γνωμοδότηση, πρόκειται για τον προσανατολισμό βάσει επιδόσεων. Το ακούσαμε πολύ και στην συζήτηση για τις απαλλαγές. Επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ και εμείς σε αυτό και στα πλαίσια του ορίζοντα του 2020 και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Πρέπει εδώ να τονίσω ότι κατά τη γνώμη μας όσον αφορά κυρίως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος τα τελευταία χρόνια. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με τις παρεμβάσεις του ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις προτεραιότητες 2020 όσον αφορά την απασχόληση κοινωνικές υποθέσεις βάσει των προκαθορισμένων στόχων. Παίρνουμε όμως πάρα πολύ στα σοβαρά τις παρατηρήσεις του ελεγκτικού συνεδρίου στην φετινή τους έκθεση και θα προσπαθήσουμε να εμπνευστούμε από τις παρατηρήσεις αυτές για να βελτιώσουμε παρετέρω τις ε, επιδόσεις στο μέλλον και την αξιολόγηση βάση επιδόσεων του προπολογισμού. Αυτά είναι τα δύο πιο σημαντικά ζητήματα που είχα να θέσω όσον αφορά τις γνωμοδοτήσεις σας. Θα δώσω το λόγο στους συναδέρφους αν θέλουν να προσθέσουν κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι, να δώσουμε το λόγο στους αδέρφους αν το επιθυμούν. Gibt es noch Bemerkungen seitens der Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τίποτα άλλο, όχι. Ούτε άλλα σχόλια έχουμε. Καλώ. Προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών 15 Δεκεμβρίου στι 12 το μεσημέρι. Παρακαλώ να το προσέξετε. 12 το μεσημέρι. Και στι 25 του μηνό θα ψηφίσουμε ενώ στην αρμόδια επιτροπή που είναι συνταγμα... ελέγχου προπολογισμού 22-23 Μάρτιο. Σημείο 9. Εγκατάσταση στη Μεσόγειο και η ανάγκη μιας κοινή προσέγγισης όσο αφορά τη μετανάστευση. Συντάκτρια γνωμοδότησής μας είναι η κυρία Ελιζαμπέτ Μαγάν Σαχτιέ. Παρακαλώ. Euh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, για την ε, έκθεση αυτή όσον αφορά την κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη μετανάστευση. Είναι μια γνωμοδότηση της Επιτροπής μας, Επιτροπής Απασχόλησης, για την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, που είναι αρμόδια επί της ουσίας. Στην ε, ΛΥΜΠΕ οι συνεισηγητές είναι η Ρομπέρτα Μέτσολα από το ΕΛΚΑ, από τη Μάλτα και ο Κασέτου Κέντζε από τους Σοσιαλιστές. Πώς προσεγγίσαμε πολιτικά την έκθεση αυτή. Επιτρέψτε μου καταρχήν να αναφερθώ στα έξι θεμέλια. Το πρώτο είναι ότι θελήσαμε να ετοιμάσουμε μία γνωμοδότηση η οποία να είναι και χρήσιμη και ρεαλιστική αλλά και συγκεκριμένη. Δεύτερον, η γνωμοδότηση αυτή πρέπει να συμπεριλαμβάνει μια από τις βασικές αρχές της Ευρώπης που είναι η αλληλεγγύη. Τρίτο σημείο. Η γνωμοδότηση αυτή πρέπει να είναι ισορροπημένη, να μην χρησιμοποιεί ακραίες θέσεις και ε, καταλήγουμε να χειριζόμαστε το προσφυγικό πολιτικά αντικά. Πρέπει να το υπενθυμίζουμε αυτό, Πρόεδρε. Τέταρτο στοιχείο. Ο πολιτικός στόχος της νομοδότησης αυτής είναι να βρεθούν λύσεις για να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα πολύ λεπτό και ευαίσθητο, αλλά πολιτικά θα έπρεπε να προσέξουμε πάρα πολύ και να αποφύγουμε κάποια πράγματα. Η ερώτηση είναι η εξής. Πώς θα εντάξουμε τους μετανάστες και τους πρόσφυγες στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας που εξακολουθεί να βρίσκεται σε κρίση. Δηλαδή, από τη μία υπάρχει η ανάγκη για αλληλεγγύη, να ενταχθούν οι πρόσφυγες κτλ. Και από την άλλη μεριά υπάρχει η πραγματικότητα της κρίσης στις ε, χώρες μας, από την οποία υποφέρουν πολλοί πολίτες μας. Πέμπτο βασικό στοιχείο. Δεν μπορούμε να πούμε απλώς ότι υποδεχόμαστε ανθρώπους χωρίς να έχουμε καμία ιδέα για το τι μπορούμε να τους προσφέρουμε. Δεν είναι θέμα αρχής, εντάξει αρχή, αλλά πέρα από την αρχή πρέπει να υπάρχει και ένα όραμα, κάτι συγκεκριμένο. Και τέλος η γνωμοδότηση αυτή λαμβάνει υπόψη τρεις κατηγορίες ανθρώπων από την μετανάστευση. Και εδώ δεν θα πρέπει να μπερδεύουμε τις κατηγορίες, γιατί υπάρχουν οι πρόσφυγες που έχουν το καθεστώς του πρόσφυγα, υπάρχουν αυτοί που ζητούν άσυλο και υπάρχουν και οικονομικοί μετανάστες. Πρόεδρε, αυτά είναι τα έξι στοιχεία στα οποία βασίστηκε ο προβληματισμός μας. Για το πρώτο, η Επιτροπή έχει εγκρίνει ένα φιλόδοξο ευρωπαϊκό θεματολόγιο και ζητάμε από το Συμβούλιο να παραμείνει στο ίδιο επίπεδο φιλοδοξίας για να υπάρχει συνοχή. Έπειτα υπενθυμίζουμε ότι μέσω πρόθεσμα το ζήτημα που θέτει το προσφυγικό και που πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη είναι το θέμα της ένταξής τους. Δεν είναι θέμα τώρα να ανοίξουμε τα σύνορα, να δεχτούμε ροές χωρίς να μπορούμε να τους εντάξουμε στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Γι' αυτό ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα σχέδιο. Ένα σχέδιο το οποίο να λαμβάνει υπόψη μια πολιτική κοινωνικής και επαγγελματική ένταξης των ατόμων αυτών. Τρίτο. Διαπιστώνουμε πόσο μεγάλη σημασία έχουν τα δεδομένα της αγοράς εργασίας. Οι μόνιμοι μηχανισμοί ε, επανεγκατάστασης. Διότι δεν πρέπει να επιδεινωθεί η πολιτική και κοινωνική κατάσταση ούτε των εδαφικών οντοτήτων, ούτε του πληθυσμού. Πρέπει να δούμε δηλαδή η ένταξη των ανθρώπων αυτών τι επιπτώσεις θα έχει επί τόπου. Και το βλέπω αυτό και από τη χώρα μου και στη δικιά μου εκλογική περιφέρεια, γιατί εκεί αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα. Τέταρτο ζήτημα, Πρόεδρε. Υπενθυμίζουμε ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι τίποτα δεν προκαταλαμβάνει την χρήση των ε, ευρωπαϊκών κονδυλίων, κυρίως του κοινωνικού ταμείου, για να συμμετέχει στην προσπάθεια ενσωμάτωσης των προσφύγων. Φυσικά μπορεί να γίνει χρηματοδότηση για την επαγγελματική ένταξη των προσφύγων. Υπενθυμίζουμε όμως ότι προσοχή Η χρήση αυτή των κονδυλίων δεν θα πρέπει από την άλλη να επιδεινώσει τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων για τους Ευρωπαίους που έχουν ανάγκη το κοινωνικό ταμείο για τη δικιά τους επαγγελματική ένταξη. Να μην δηλαδή σε βάρος όλων των πολιτικών μας για την ένταξη των νέων, για την ένταξη των γυναικών, των ηλικιωμένων κλπ. Πέμπτον, ζητάμε από την Επιτροπή σε συνεννόηση με τα κράτη-μέλη να καταρτήσει ένα σύστημα για την επιτάχυση των διαδικασιών για την ισοτιμία των διπλωμάτων και την αναγνώριση δεξιοτήτων. Έχουμε να κάνουμε με πληθυσμό προσφύγων που είναι μορφωμένοι αλλού, σε άλλες χώρες βέβαια, με άλλα συστήματα μόρφωσης και εκπαίδευσης. Δεν μπορεί να υπάρξει ένταξη αν δεν υπάρξει αναγνώριση των διπλωμάτων τους και αν δεν υπάρχει αυτή η πολιτική γρήγορης ένταξής τους. Έκτον, προειδοποιούμε την Επιτροπή για το κίνδυνο που υπάρχει από την παράνομη εργασία των μεταναστών. Πρέπει να είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι για τις κυρώσεις που προβλέπονται κατά των εργοδοτών εκείνων οι οποίοι θα απασχολούσαν μετανάστες στα πλαίσια της οδηγίας των εποχιακών εργαζόμενων. Υπάρχουν κυρώσεις, αλλά πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε ένα καλύτερο ακόμα σύστημα. Τέλος. Είναι πολύ σημαντικό να επενθυμίσουμε τους κινδύνους τόσο για τον εργαζόμενο όσο και τον εργοδότη από την υπογραφή σύμβασης εργασίας ενός ετούντα άσυλο στην περίπτωση που η αίτηση παροχή ασύλου απορριφθεί. Αυτό ε, έθετε, θα σε κίνδυνο όλες τις πλευρές. Πρέπει να είμαστε λοιπόν προσεκτικοί και να προβλέψουμε όλες αυτές τις περιπτώσεις εκ των προτέρων. Τέλος, ζητάμε από την Επιτροπή να είναι φιλόδοξη όσον αφορά την οδηγία για την μπλε κάρτα, ώστε να αυξηθεί η προβολή της και η αποτελεσματικότητά της και να προσελκύσει εργατικό δυναμικό υψηλής ειδίκευσης. Ένα τέτοιο εργατικό δυναμικό θα μπορούσε να προσφέρει στην Ευρώπη πολλά ωφέλη. Αυτά λοιπόν είναι τα θέματα πάνω στα οποία βασιστήκαμε για να εκπονήσουμε τη γνωμοδότηση αυτή. Το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή τροπολογιών είναι 15 Δεκεμβρίου. Μας συμφέρει να δουλέψουμε μαζί, να συνεργαστούμε, ώστε αυτή η πρώτη βάση εργασίας που έχουμε να προχωρήσει από κοινού. Εγώ ευχαρίστω συνεργάζομαι με όλους τους σκιώδεις εισηγητές από όλες τις πολιτικές ομάδες. Ελπίζω τόσο για την έκθεση αυτή, την ονομαδότηση αυτή, όσο και για άλλες που ψηφίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, θα έχουμε επικοδομητικές συζητήσεις και θα δείξουμε ότι η Επιτροπή Απασχόλησης είναι σε θέση να πετύχει συνενέσεις και να ξεπεράσει προβλήματα τα οποία μας διχάζουν. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να προωθήσουμε μια πραγματική πολιτική στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαι στη διάθεσή σας τώρα και στη διάθεση όλων των πολιτικών ομάδων για να συνεργαστούμε με θετικό πνεύμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. So, dann hat Xavi Ο Χάβι Λόπεθ Φερνάντες έχει το λόγο, αλλά θα πρέπει να θυμίσω ότι από χρόνο δεν πάμε πολύ καλά. 20 λεπτά για κάθε θέμα έχουμε υπολογίσει, αλλά πρέπει να μιλάμε λίγο πιο γρήγορα. Για κάθε item έχουμε ένα 20 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τις εξηγήσεις σας, ε, για την ε, προοπτική που σε πολύ μεγάλο βαθμό συμμεριζόμαστε και θέλω να πω ότι είναι από τις μεγαλύτερες προκλήσεις ε, του ευρωπαϊκού εγχειρήματος αυτή τη στιγμή. Και καλό είναι να γνωμοδοτεί και η δική μας Επιτροπή από τη δική μας σκοπιά προφανώς. Μιλάμε εμείς για την ένταξη στην αγορά εργασίας. Συμφωνώ με την εισηγήτρια για τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τα πράγματα και τι έχουν συμβεί τους τελευταίους μήνες. Δυστυχώς υπήρξε η αίσθηση ότι δεν δόθηκε αρκετή απάντηση, αρκετές απαντήσεις στα προβλήματα με τα οποία ασχολούμαστε μεν, αλλά όχι επαρκώς. Αν σταθούμε λίγο να δούμε τι συζητήσαμε, πραγματικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ένα φιλόδοξο ρόλο, ε, κατέθεσε προτάσεις και πολλές φορές το Συμβούλιο ήταν εκείνο το οποίο δεν εστάθη στο ύψος των περιστάσεων, γιατί είναι πολύ κρίσιμη στιγμή και σοβαρή. Είχαμε περίπου ένα εκατομμύριο φίξεις, έτσι δεν είναι πάρα πολύ γρήγορα ε, τη διάρκεια του έτους. Αυτή είναι λοιπόν η σκοπιά και η προοπτική και συμφωνούμε με τη γνωμοδότηση. Προφανώς θα πρέπει να το συζητήσουμε εδώ στην Επιτροπή μας και να εξηγήσουμε με κάθε ειλικρίνεια ότι αυτό που οφείλουμε να κάνουμε ως διεθνής κοινότητα και ως Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, να αναλάβουμε τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά μας από τη Σύμβαση της Γενέβης και εκείνοι που έχουν δικαίωμα στο άσυλο να βρίσκουν και προστασία κάπου στην Ευρώπη και να μην υπάρχουν δυσκολίες και εμπόδια για την ένταξή τους και την κοινωνική και την εργασιακή. Βεβαίως θα πρέπει να γίνει μια κοινή προσπάθεια με ευελιξία, με έξυπνες δημόσιες πολιτικές προς την κατεύθυνση αυτή. Για όλα αυτά λοιπόν υποστηρίζω γενικά και η ομάδα μου, τα όσα είπε η συντάκτρια, ελπίζω να ανταλλάξουμε και απόψεις για να βελτιώσουμε λίγο ε, την γνωμοδότηση. Απλώς να προσθέσω δύο-τρία πράγματα. Προσοχή από πού θα βρούμε τα λεφτά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Στην πρόταση που μας κάνετε δεν λέει τίποτα που να αποκλείει ότι θα φύγουν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Εμείς όμως έχουμε εξηγήσει 100 φορές ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε χρήματα από το Κοινωνικό Ταμείο που θα βρουμε τα λεφτα ειναι πολυ σημαντικο αυτο στην προταση που μας κανετε δεν λεει τιποτα που να αποκλειει οτι θα φυγουν απο το ευρωπαικο κοινωνικο ταμειο εμεις ομως εχουμε εξηγησει 100 φορες οτι δεν μπορουμε να βγαλουμε χρηματα απο το κοινωνικο ταμειο που θα πηγαινε στους πιο ευάλωτους της κοινωνίας για να τα δώσουμε στους πρόσφυγες. Είναι πολύ ευαίσθητο αυτό το θέμα και λεπτό. Συμφωνώ με την ιδέα από τη μια να προσπαθήσουμε να καταπολεμήσουμε τους εξτρεμισμούς. Το πρόβλημα όμως ποιο είναι. Εάν με καλές προθέσεις, δεν λέω, παίρνουμε λεφτά από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες, αλλά δεν βάζουμε επιπλέον χρήματα, τελικά τι θα κάνουμε. Βάζουμε ένα κοινωνικό αυτοματισμό και ε, έναν ανταγωνισμό των προσφύγων με τους ανθρώπους που είναι πάμφτωχοι. Και αυτό είναι νερό στο μήλο της ακροδεξιάς. Ας είμαστε ξεκάθαροι και ειλικρινεί Να δούμε από πού θα βγουν τα λεφτά και να μην βάζουμε σε ανταγωνισμό ή σε σύγκρουση τους πιο φτωχούς της κοινωνίας με τους πρόσφυγες. Είναι πολύ σημαντικό να ενταχθούν στον εργασιακό βίο. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να κάνουμε και μηχανισμοί, ας πούμε, να τους μάθουμε τι γλώσσες, δεξιότητες κτλ. Υπάρχουν δυνατότητες, αλλά κατά την άποψή μας, η γνωμοδότηση της Επιτροπής της δικής μας κοινωνικών θεμάτων και απασχόλησης θα είναι από τις σημαντικότερες στη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκέρικε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια Μωράν Σαχτιέ για την πρόταση της νομοδότησης. Εγώ είμαι Γερμανός Ευρωβουλευτής και την υποστηρίζω απολύτως όταν ζητάει να εφαρμόζονται ε, ε, όσα ορίζει το θεματολόγιο για τη μετανάστευση. Θα πρέπει να σταματήσει η εμπλοκή στο Συμβούλιο. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίζει εκείνους που έχουν αναγνωριστεί ως ε, πρόσφυγες και ε, όποιος ως ε, χώρα κάνει περισσότερα θα πρέπει να παίρνει και χρήματα και όποιος δεν θέλει να κάνει τίποτα θα πρέπει να πληρώνει. Ε, και είμαστε και υπέρ της απασχόλησης αλλά προσοχή στη διατύπωση. Δεν είναι ο κάθε μετανάστης πρόσφυγας, ούτε ο κάθε πρόσφυγας είναι μετανάστης. Ας κάνουμε αυτή τη διάκριση. Αλλιώς πώς να καταλάβουν οι πολίτες τι γίνεται. Στόχος ποιος πρέπει να είναι. Να επιτραπεί σε πολλούς η ταχεία επιστροφή στις πατρίδες τους. Εδώ συζητούμε την ιδιαίτερη κατάσταση στη Μεσόγειο και θέλω να πω τα εξή ζητήματα. Τρία. Πρώτον, κάθε οικογένεια προσφύγων που δεν πέφτει στα νύχια των ε, διακινητών και δεν κινδυνεύει να σκύλο πνιγεί είναι ε, ένα κέρδος για την ανθρωπότητα. Θα πρέπει να σταθεροποιηθούν οι περιοχές από τις οποίες προέρχονται οι άνθρωποι αυτοί για να μην πηγαίνουν στη θάλασσα. Δεύτερον, το Ισλαμικό κράτος ε, απειλεί περιοχές της Συρίας. Ε, πριν από τέσσερις εβδομάδες εγώ είχα πάει στην Ιορδανία σε ένα καταβλησμό προσφύγων και ματώνει η καρδιά μου γιατί ένα κοριτσάκι που γεννήθηκε στο Ιράκ και μεγαλώνει εκεί στο καταβλησμό και θέλει να γίνει γιατρό, σαν τη μαμά τη. Αλλά πώ θα μπορέσει. Ε, πρέπει εμεί να δώσουμε αυτές τις ευκαιρίες αυτά τα παιδιά να μορφωθούν. Και ένα τελευταίο, το Ισλαμικό κράτο στην Αφρική. Παράλληλα ε, με εμά συνεδριάζει η αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΚΕ. Και πολλοί συνάδελφοι μου λένε ότι εκεί γίνεται μια ανίερη συμμαχία Ισλαμικό κράτο και Μπόκο Χαράμ στη Βόρεια Αφρική. Θα πρέπει λοιπόν να το έχουμε υπόψη μας αυτό γιατί όταν συζητούμε για τη Μεσόγειο έχουν σημασία αυτά τα θέματα και χρειάζεται ένας πιο ενεργός ρόλος της ε, Ένωσης για τη Μεσόγειο που μάλλον αδρανεί. Χρειάζεται μεγαλύτερη δράση σε συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση. Ας δράσουμε επιτέλους. Ευχαριστώ πολύ. Ο Καλβέ Σαμπόμ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω στα γαλλικά και θα μιλήσω και ισπανικά, αλλά αρκετά σύντομα. Πρώτα απ' όλα στα γαλλικά για να απαντήσω και στα σχόλια της κυρίας Μωρά Σαρτσέ. Διότι εκείνη μας ε, απέστειλε τα πρώτα μηνύματα μιλώντας για, τις μεγάλες, ε, για τα μεγάλα επιτέγματα της περασμένης εβδομάδας, τη μεγάλη συμφωνία, αλλά Υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις ψευδοπολιτικών, οπότε δεν είναι ανάγκη να είμαστε περήφανοι για όλα αυτά. Ε, αυτά που προτείνει η κυρία Μωράν Σαρτιέ μου φαίνονται κάπως αυτονόητα ε, οπότε, και η ομάδα της προτείνει, οπότε πώς να μην τα κανείς, είναι μια πολύ καλή βάση εργασίας που θα μπορούσε κανείς ε, ευθύς εξ να την αποδεχτεί. Από τη δική μας πλευρά, τη δική μου δηλαδή. Θα πρότεινα κάποιες γλωσσικές βελτιώσεις, γι' αυτό και μιλώ στα γαλλικά, ίσως είναι θέμα γαλλικής γλώσσας, δηλαδή να ε, προωθηθεί η διάθεση, το πρόβλημα των προσφύγων που θα έρθουν στην Ευρώπη δηλαδή, είναι το θέμα η ένταξή τους στην ευρωπαϊκή κοινωνία, λέει. Ε, να προσέξουμε ότι πρέπει να μιλάμε για πρόσφυγες και όχι μετανάστες και το θέμα είναι και δική τους βούληση για ένταξη. Η μεγάλη διαφορά μεταξύ πρόσφυγα και μετανάστη είναι ότι συνήθω ο πρόσφυγα θέλει να γυρίσει κάποια στιγμή στην χώρα του όταν ε, οι συνθήκε δημοκρατικέ επιστρέψουν, όταν υπάρχουν συνθήκε κανονικέ διαβίωση, όταν επιστρέψουν οι γιατροί, οι αρχιτέκτονε και το καθεξή. Και πέραν αυτού, ξέρουμε ότι υπάρχει μετανάστευση από την Ασία λόγω χάρη που ποτέ δεν είχε πρόβλημα ένταξης. Να φροντίσουμε λοιπόν εδώ να είμαστε κάπως προσεκτικοί. Ε, κοινωνικές πολιτικές για την ένταξη, ναι, αλλά και η επαγγελματική στήριξη μπορεί να ε, δώσει αυτή τη διάθεση για ένταξη. Δεύτερο σημείο, όταν να προειδοποιούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον κίνδυνο της παράνομης εργασίας, ο κίνδυνος ως έκφραση στις μέρες μας είναι κάπως ε, ιδιαίτερος όρος. Δηλαδή, κινδύνο μπορεί να είναι κανεί να μια μπύρα σε μια τεράστια στο Παρίσι, λόγω χάρη. Είναι μια πραγματικότητα αυτό ο κίνδυνο που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, όπω η παράνομη εργασία για κάποιε περιπτώσει. σω λοιπόν ο όρο κίνδυνο να άλλαζε με στρέβλωση ή με μεγάλη έλλειψη ισορροπία που έχει προκληθεί. Και τώρα θα μιλήσω ισπανικά. Ε, όπω και προλαλή σα. Θα είμαι σύντομο όταν θα έχω τελειώσει με τα γλωσσικά. Λοιπόν, ισπανικά. Συνεχίζει στα ισπανικά, βάλτε τα ακουστικά σας, λέω μιλητή κλπ. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και συμφωνώ με τον κύριο Λόπε, τον Θαβίδη Λόπε. τον συναδελφό μου, να είμαστε προσεκτικοί με τα κονδύλια και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Γιατί έχουμε μια, έναν προπολογισμό αντιευρωπαϊκό. Αν προσπαθούμε να τα κάνουμε όλα με αυτόν τον προπολογισμό, ε, δεν θα τα καταφέρουμε. Να είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί και να βάζουμε προτεραιότητες. Αν θέλουμε πραγματικά, ας βάλουμε μια ειδική γραμμή για την μετανάστευση ή ένα ειδικό ταμείο ή υποταμείο αλλά να ξέρουμε τι βάζουμε εκεί. Για να μην υπάρχει αντιπαράθεση τι θα πάρουμε από αυτή τη γραμμή και θα πάρουμε από την άλλη γραμμή, για ποιο σκοπό από τη μία και ποιο σκοπό από την άλλη. Έπειτα, να διαχωρίσουμε πολύ καλά το ποιο είναι μετανάστης και ποιο είναι πρόσφυγας. Έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Στη Θέοτα και Μελίγια το είδαμε εμείς. Δημιουργείται διαφορετική προβληματική στιγμή και την άλλη περίπτωση. Ένα γιατρό που έχει φύγει, είναι πρόσφυγας και θέλει να ξαναγυρίσει στη χώρα του να δουλέψει πάλι εκεί γιατρός, είναι κάτι εντελώ διαφορετικό από ένα μετανάστη ο οποίο θέλει να εγκατασταθεί στην Ευρώπη για να βρει δουλειά στην Ευρώπη και να μείνει μονίμω εκεί. Δύο πράγματα μου λείπουν εμένα εδώ. Το ένα είναι. Α δούμε τον τίτλο. Τι λέει ο τίτλο. Λέει η κατάσταση στην περιοχή της και η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη μετανάστευση. Ε, συμφωνώ και είναι πολύ ενδιαφέρον. Και ακριβώς εδώ είναι που πρέπει να ξυπνήσει το Συμβούλιο και να ακούσει αυτά που λέμε. Αλλά από πλευρά της απασχόλησης ένα θέμα που έχει να κάνει με μια ολιστική προσέγγιση απαιτεί και κάτι θετικό. Θετικό πρώτον όσον αφορά τις ανάγκες της συνολικής μας αγοράς εργασίας στην Ευρώπη. Και αναπόφευκτα είναι κάτι πάνω στο οποίο έχω δουλέψει για πολύ καιρό εγώ. Αν δούμε ολιστικά τη μετανάστευση, η οποία γίνεται με βούληση, ε, συντεταγμένα, τότε αυτή η ολιστική πολιτική πρέπει να λάβει υπόψη και τα σοβαρά δημογραφικά προβλήματα που έχουμε στην Ευρώπη και που δεν είναι τα ίδια σε όλες τις χώρες. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Σε άλλες χώρες όπως η δικιά σας ή η δικιά μου πρόεδρο υποφέρουν. Λοιπόν, θα έλεγα, αν μη τι άλλο, να συμπεριλάβουμε στην γνωμοδότηση αυτή ότι ένα ολιστικό πρόγραμμα για την ε, μετανάστευση πρέπει να λάβει υπόψη και την αγορά εργασίας την ευρωπαϊκή, αλλά και το δημογραφικό γιατί πρέπει να δούμε ποιος είναι ο αντίκτυπος, τα προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης κλπ. κλπ, κλπ. Ευχαριστώ. Ο Πατρίκ Λιουγιαρίκ κανονικά έχει το λόγο, αλλά απουσιάζει. Οπότε η Τζιν Λάμπερτ, η οποία έχει ζητήσει συγγνώμη γραπτός, γιατί είναι σε άλλη συνεδρίαση και κολλείται. οπότε είναι εντάξει, δικαιολογημένος απούσα. Η κυρία Ατζέα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια, την κυρία Μωράν Σαρτιέ. Βεβαίω και θα συνεργαστούμε με κάθε παρέτη προθυμία και απλώς να επισημάνω κάποια σημεία επικριτικής τοποθέτησης. Θέλουμε μια ολιστική προσέγγιση και βλέπουμε ότι αυτή η κοινή προσέγγιση είναι κάτι που απαιτείται. Είναι η μόνη δυνατότητα για να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα σε μια πραγματικότητα που διαρκώς μας προλαμβάνει. Η σύνοδος της Βαλέτα, της Λαβαλέτα, έδειξε μια σαφή ένδειξη για το πώς πρέπει να χειριστούμε το θέμα της μετανάστευσης και δύο μέρες μετά ε, πολλές χώρες έκαναν ακριβώς τα αντίθετα από όσα συζητήθηκαν. Καταλαβαίνω λοιπόν Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά το πρόβλημα. Καταλαβαίνω γιατί λήφθησαν κάποιες αποφάσεις από ορισμένου. Όμως δεν μπορούμε να λέμε κάτι και την επόμενη μέρα να βάζουμε σειρματοπλέγματα ή να υψώνουμε τύχη. Διότι είτε την ολιστική προσέγγιση την ελαμβάνονται 28 χώρε είτε μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Χαίρομαι Ιδιαίτερα που η συνάδελφος μιλά για ε, μεσοπρόθεσμη προσέγγιση, διότι αυτό δείχνει ότι χρειάζεται ένα πρόγραμμα με κάποια σχετική διορατικότητα. Αλλά θα θέλαμε να δούμε και την ανάγκη μιας άμεσης αντίδρασης. Υπάρχει ένα πρόβλημα έκτακτο και η αδυναμία μας να χειριστούμε τις κατεπίγουσες συνθήκε Έχουμε έναν καταμερισμό 200.000 προσφύγων και την πράξη λιγότεροι από 200 έχουν μετατοπιστεί. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε μη αποτελεσματικοί. Περιμένω λοιπόν αυτή η απαραίτητη θεώρηση και το επαναλαμβάνω. Χαίρομαι ιδιαίτερω που έχει δοθεί αυτή η διάσταση τη μεσοπρόθεσμη προσέγγιση. Πρέπει όμω να δούμε και τι έκτακτε ανάγκε που έχουμε τώρα να αντιμετωπίσουμε. Χρήση των κονδυλίων. Πολλές είναι οι ευρωπαϊκές χώρες που δεν ε, έχουν καλά αποτελέσματα στη χρήση των κονδυλίων και σε ό,τι αφορά τη χώρα τους κιόλα. Ή θα αλλάξουμε την προσέγγιση μας και θα πετούμε ορθολογιστική χρήση και αποτελεσματική εκτέλεση των κονδυλίων με παρακολούθηση πολύ προσεκτική στη χρήση αυτών ή εφόσον πρέπει να συμπεριλάβουμε να εντάξουμε και άλλες δυνατότητες χρήσης για την ένταξη στον χώρο εργασίας και στις κοινωνίες μας των μεταναστών, τότε θα χαθούμε σε ένα ε, τέλμα. Ένα τέλμα, ένα βάλτο που δεν θα ξεφύγουμε ποτέ το ελεγκτικό συνέδριο συνεχίζει να μας ε, επιτιμά ή τέλος πάντων να μας επικρίνει ότι δεν είμαστε αποτελεσματικοί, ότι δεν πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Φανταστείτε τι θα γίνει εάν η ψαλίδα ε, για την κακή χρήση των κοντιλίων αυτών μεγαλώσει κι άλλο. Κάτι άλλο που θέλω να τονίσω είναι τα γλωσσικά μαθήματα για να μπορέσουν να ενταχθούν αυτά τα άτομα, καθώς και ο ρόλος όσων θα αναλάβουν την εκπαίδευση στα σχολεία στους τόπους μάθησης. Κάποιε φορέ δεν καταφέρνουμε ούτε να αναγνωρίσουμε, να έχουμε αποτελεσματική αναγνώριση των μεταναστών. Εγώ είμαι Ιταλίδα. Έχουμε τρία hot spot, τρία σημεία υποδοχή, όπου θα έπρεπε να γίνεται η ταυτοποίηση των μεταναστών. Και εμεί θέλουμε να μάθουν και τη γλώσσα, αλλά ακόμα δεν μπορούμε καν να του ταυτοποιήσουμε. Ε, εδώ λοιπόν Νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρές αυτές οι ενδείξεις που έχει καταγράψει η συνάδελφος, αλλά έχουμε προβλήματα άμεσης ανάγκης, πολύ σοβαρά, που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και σε επίπεδο Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων έχουμε και εκεί πολλές υποχρεώσεις, διότι εάν θέλουμε να ακολουθήσουμε τον δρόμο της ένταξη, θα πρέπει να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της ε, ένταξη αυτής. Θα πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί. Εκεί που θέλουμε πραγματικά να ενταχθούν αυτοί οι άνθρωποι, θα πρέπει να του εγγυηθούμε ελάχιστα πρότυπα σεβασμού εργαζομένων που εντάσσονται προ ένταξη, αλλά και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολλέ φορέ ούτε τα, ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών δεν καταφέρνουμε να σεβαστούμε. Πέραν αυτού και πέραν των δικών μου προσωπικών παρατηρήσεων, με κάθε χαρά θα συνεργαστούμε για τη σύνταξη αυτού του κειμένου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λίγα λόγια διότι εφόσον μιλάμε πάλι για μετανάστευση, να πω ότι στην Ιταλία εντωμεταξύ έρχονται χιλιάδες μετανάστες. Δεν έρχονται λαθρέα. Διότι είναι παράνομοι αυτοί που έρχονται στην Ιταλία. Στην Ιταλία, λοιπόν, είναι πρόσφυγες οικονομικοί μετανάστες, κάποιοι εγκληματίες, όταν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την αναγνώριση του καθεστώτος ε, πρόσφυγα. Αυτές, αυτά τα άτομα λοιπόν 1,5 χρόνο κυκλοφορούν ελεύθερα στη χώρα μας. Κάποιοι ε, εργάζονται στη μαύρη αγορά, κάποιοι παραμένουν σε κάποιο ξενοδοχείο εις βάρος της δικής μας κοινωνίας. Αυτό προφανώς δημιουργεί κοινωνικές εντάσεις, διαρκή κοινωνική ένταση. Δεν θα ήθελα λοιπόν εδώ απλώς να συζητούμε ε, για πολλωστή φορά μια έκθεση, για πολλωστή φορά μία ε, θεωρητική σκέψη με περιττά λόγια, με άδειε κουβέντε. Διότι όσο συζητάμε η κατάσταση επιδεινώνεται και η Ευρώπη δεν ήθελε να λάβει γνώση, δεν ήθελε να αντιμετωπίσει πριν από κάποια χρόνια το πρόβλημα τη μετανάστευση. Σήμερα βρισκόμαστε απροετοίμαστοι και πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Σημειώνω την ε, προθυμία του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ε, ασχοληθούν επιτέλους με το θέμα σοβαρά. Το Κοινοβούλιο όμως το έχει συζητήσει Ε, Λίγο πολύ είχαμε όλοι πει ότι έχουμε την πεποίθηση ότι το θέμα της μετανάστευσης και της κοινωνικής ένταξης των προσφύγων πρέπει να αντιμετωπιστεί, αλλά βλέπω στην Ιταλία η κατάσταση διαρκώς να επιδεινώνεται. Όλο και χειρότερα. Ε, και μια απάντηση σε έναν συνάδελφο που κάτι σχολίασε προηγουμένως. θα έλεγα ότι δεν μπορεί να. Θα έλεγε κανεί ότι δεν μπορεί κανεί να ασχολείται με μετανάστευση, ένα πολιτικό τη ακροδεξιά. Εγώ δεν είμαι ούτε τη ακροδεξιά ούτε τη δεξιά. Είμαι απλώ ε, πολιτικό που είναι πολύ προσεκτική ε, και κοιτάζει με μεγάλο ενδιαφέρον όσα συμβαίνουν στη χώρα του. Ε, και η χώρα μα, οι Ιταλοί και οι Ιταλίδε ζητούν από την Ευρώπη να αντιμετωπίσουμε με σοβαρό τρόπο το θέμα τη μετανάστευση. Πέραν λοιπόν των ωραίων λόγων που σήμερα μπορούμε να εκφωνούμε, ε, θα πρέπει να είμαστε πιο τολμηροί, πιο αποφασιστικοί και στο Ευρωκοινοβούλιο, διότι δεν μπορούμε να επιτρέπουμε στους εαυτούς μας ε, να συνεχίζουμε επί μήνες και επί χρόνια να συντάσσουμε απλώς εκθέσεις. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε στους εαυτούς μας να περιμένουμε το επόμενο, την επόμενη σύνοδο κορυφής για τη μετανάστευση, την επόμενη έκτακτη σύνοδο για την μετανάστευση, διότι καθημερινά φτάνουν στις ακτές μας, στη χώρα μας, άτομα που κάποια χρειάζονται βοήθεια. Κάποιοι έρχονται απλώς μέχρι να διαπιστωθεί η ταυτότητά τους και να βρεθεί και το κουράγιο να τους ξαναστείλουμε στην χώρα τους. Πρέπει λοιπόν και με αυτό να ασχοληθούμε. Υπάρχουν κάποια άτομα που φτάνουν και έχουν δικαίωμα να έχουν το καθεστώ του πρόσφυγα και χρήζουν αρρωγή, κάποιοι όμω πρέπει να γυρίσουν σπίτι του. Αυτό δυστυχώ δεν γίνεται ακόμη. Και αυτό δημιουργεί διαρκώ κοινωνικέ εντάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη μα. Ο πρόεδρος, η κυρία Χέλγα Στίβενς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε και συνάδελφοι. Ο σκιώδης εισηγήτρια της ΕΣΙΑ ε, για την έκθεση ε, στην ΛΥΜΠΕ και στην ΕΜΚΟ έχω μια βασική ε, παρατήρηση να κάνω. Προηγουμένως όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συντάκτρια της νομοδότησης για την ενημέρωση και για την ε, εξαιρετική της δουλειά και τη συνεισφορά της με το κείμενο. Οι παρατηρήσεις μου τώρα. Θέλω να τροποποιήσω τη δεύτερη παράγραφο της νομοδότησης όπως προτείνεται γιατί θέλω πολύ πιο συγκεκριμένα να τα λέει αυτά και να διευκρινίζει. Τι εννοώ. Θα πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει χρήση του δικαιώματος πρωτοβουλίας για να τροποποιηθεί η οδηγία ε, για ε, τα προσόντα ε, και να προσαρμοστεί στην Σύμβαση Γενέβης του 1951. Από την πρώτη μέρα ο πρόσφυγας έχει τα ίδια δικαιώματα με τους γηγενείς αυτόχθονες που όλη τους τη ζωή έχουν εργαστεί για ε, τα δικαιώματά τους. Ο Βέλγιο αυτό έχει δημιουργήσει κάποια δυσφορία στον πληθυσμό ε, όταν γίνεται για αναδιανομή και ανακατανομή των προσφύγων. Ε, και αυτό που έχει σημασία ή των ετούν τον άσυλο. Επίσης, το θέμα της ανεργίας. Ποιος ετών άσυλο που κέρδιζε 600 ευρώ Ε, θα δουλέψει όταν του δίνουν επίδομα 3.000 με το καλημέρα σας για όλη την οικογένεια. Γιατί να πάει να δουλέψει. Λοιπόν, το δικό μου μήνυμα ποιο είναι. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ας κάνουν τη δική τους πολιτική ένταξης. Γι' αυτό η οδηγία για τα προσόντα και τις δεξιότητες θα πρέπει να ε, βρίσκει μια πιο ελαστική εφαρμογή όπως προβλέπει και η Σύμβαση για τους Πρόσφυγες. Θα κάνω λοιπόν τροπολογία, σας ζητώ να την υποστηρίξετε και θα σας στείλω το συντομότερο το σχετικό κείμενο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η Αγνιέσκα Κοσλόσκα Χαράγεβιτς, αν το λέω σωστά το όνομά σας. Ε, ε, ευχαριστώ. Συγχαρητήρια, Ελίζαμπετ. Ευχαριστούμε για αυτή, στο τον εξαίρετο ορισμό και για τόσα λες για την πολιτική απέναντι στην μετανάστευση. Και ευχαριστώ που έλαβες υπόψη σου και τον έλεγχο και την ένταξη. Δεδομένης της κλίμακας του φαινομένου, είναι πολύ σημαντικό όσο γίνεται πιο γρήγορα να μπορέσουμε να εντάξουμε τους μετανάστες που θέλουμε να εντάξουμε τους οικονομικούς για να αρχίσουν να δουλεύουν. Το σημείο 5 είναι ισοτική σημασία γιατί αναφέρεται στην επιτάχυνση των διαδικασιών για την ισοτιμία των διπλωμάτων, για την αναγνώριση δεξιοτήτων. Μερικέ φορέ η διαδικασία αυτή κρατάει χρόνια. Όταν έρχεται στη χώρα μα ένα γιατρό και περιμένει 6 χρόνια για να αναγνωριστεί το δίπλωμά του, καταλαβαίνετε ότι και χρόνο χάνει, αλλά ξεχνάει για τη δουλειά του. Δεν έχει νόημα πια. Ενώ είναι κάποιος ο οποίος θα μπορούσε κάλλιστα να δουλέψει. Οπότε και ο ίδιος είναι πολύ απογοητευμένος και από την άλλη μεριά και η οικογένειά του πλήττεται γιατί δεν μπορεί να υποφεληθεί. Γι' αυτό και θα έπρεπε όσο γίνεται πιο γρήγορα να φροντίσουμε για την οικονομική ανεξαρτησία των ανθρώπων αυτών. Η αναγνώριση δεξιοτήτων είναι ένα ζήτημα που έχει σημασία και μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Και εκεί υπάρχει κόλλημα ακόμα. Όλα όσα αναφέρονται στην ένταξη τώρα πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικά. Εννοείται ότι η ένταξη ενσωμάτωση αυτή περνάει από την εκπαίδευση των νέων, των ενηλίκων κτλ. Ε, να μαθαίνουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής και όσον αφορά τον έλεγχο τώρα, οι άνθρωποι εκείνοι που είναι παράτυποι, ξέρουμε ότι τα δύο τρίτα εκείνων που δεν θα πάρουν άσυλο θα παραμείνουν στη χώρα. Όλο και περισσότεροι δε. Οπότε συσσωρεύονται. Κάθε μήνας που περνάει, κάθε εξάμηνο, από ό,τι φαίνεται είναι όλο και περισσότεροι αυτοί που μένουν. Πολύ σύντομα λοιπόν ο αριθμός των παράνομων αυτών μεταναστών ε, θα κάνουν και παιδιά. Που δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και στη μόρφωση. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλος κίνδυνος είναι κάτι τέτοιο. Ακόμα και αν αυτά τα παιδιά γεννηθούν και μεγαλώσουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρόβλημα θα είναι τεράστιο. Και δεν πρόκειται μόνο για την ευημερία των ανθρώπων αυτών που ζουν δίπλα μας, αλλά πρόκειται και για την ασφάλειά τους. Και όχι μόνο τη δική τους, αλλά και τη δική μας. Πολύ σημαντικό. Τέλος, έρχομαι στην αναθεώρηση της οδηγίας για την μπλε κάρτα και για την παράνομη εργασία. Πολύ συχνά την προβληματική αυτή την ξεχνάμε στη συζήτηση. Πάρα πολλοί άνθρωποι φτάνουν παράνομα στην Ευρώπη, ενώ θα μπορούσαν νομικά, νόμιμα, ε, να το κάνουν, να έρθουν και να δουλέψουν και να βοηθήσουν και στην ανάπτυξη ευρωπαϊκής οικονομίας. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι για όλες αυτές τις προτάσεις σας, οι οποίες πιστεύω ότι είναι σωστές. Ευχαριστώ. Κωνσταντίν κυρία Κούνεβα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ την καλή συνάδελφο κυρία Μωρίν Σαρτία την πάντα καλή δουλειά που κάνει. Ωστόσο έχω κάποιε παρατηρήσει όσον αφορά την γνωμοδότησή τη. Φοβάμαι πώ δεν υπάρχει κάποιο πραγματικό φιλόδοξο σχέδιο από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τη μετανάστευση και φυσικά ούτε και από την πλευρά του Συμβουλίου. Επιπλέον το τελευταίο διάστημα που κάποιοι έχουν συνδέσει την τρομοκρατία με τη μετανάστευση, κάποια κράτη-μέλη δυστυχώ έχουν βρει αφορμή να κλείνουν τα σύνορά του και να αφήνουν όλο το βάρο στο νότο τη Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα. Για να μιλάμε για πραγματικά μέτρα που θα βοηθήσουν τους μετανάστες να ενσωματωθούν, πρέπει να μιλήσουμε πρώτα για ισότιμη κατανομή των μεταναστών Όσο δεν το κάνουμε αυτό, πώς θα μιλάμε για μέτρα αποτελεσματικής αντιμετωπίσης και ενσωματώσεις. Σε ποια κοινωνία, με ποιο εργασιακό προγραμματισμό τα, ε, τα μπορούσαμε πολλά να κάνουμε και όσον αφορά τη ζήτηση και την προσφορά αν δεν λύσουμε τα βασικά προβλήματα θα λειτουργούμε πρόχειρα και πυροσβεστικά. Χρειάζεται πολύ καλός προγραμματισμός για το τι αντέχει και το τι οφείλεται να προσφέρει κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας θυμηθούμε επιτέλους ουσιαστικά την αρχή της αλληλεγγύης της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φοντούλης, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, η Ευρώπη θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τι θέλει. Ο πρόεδρος Γιούγκερ ζητούσε 50 εκατομμύρια μετανάστες επειδή η Ευρώπη γερνάει. Αλληλεγγύη ναι, ανθρωπισμός ναι. Αλλά η πολιτική των ανοιχτών συνόρων γύρισε μπούμεραν στην Ευρώπη. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν είναι όλοι οι μετανάστες πρόσφυγες. Η πλειοψηφία τους είναι οικονομικοί μετανάστες που αναζητούν μια καλύτερη ζωή. Είναι θεμητό. Κάθε άνθρωπος να αναζητά μια καλύτερη διαβίωση για αυτόν και την οικογένειά του. Μετά την πρόσκληση που έκανε η Ευρώπη σε αυτούς τους ανθρώπους, όταν είδε τις ορδές των μεταναστών και τη διείσδυση ανάμεσά τους τρομοκρατικών στοιχείων με τα γνωστά αποτελέσματα, έκλεισαν τα σύνορά τους. Και όλοι αποποιούνται των ευθυνών τους. Φταίει η Ελλάδα για την αθρώα προσέλευση μεταναστών. Εάν η Ελλάδα δεν έδειχνε την ευαισθησία να διασώζει καθημερινά εκατοντάδε ζωών στα νερά του Αιγαίου, τι θα λέγανε στην Ευρώπη, ότι δεν σέβεται την ανθρώπινη ζωή και βουλιάζει τις βάρκες με τους μετανάστες. Τώρα τι λένε οι Ευρωπαίοι, ότι τα σύνορα της Ελλάδας δεν φυλάσσονται, ότι είναι τρύπια σαν ελβετικό τυρί και περνάνε οι χιλιάδες μετανάστες προς την Ευρώπη. Σας ερωτώ, εάν όλοι αυτοί οι άνθρωποι με το κλείσιμο των συνόρων μείνουν εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα, πώς θα επιβιώσουν όταν δεν υπάρχουν δουλειές και η ανεργία είναι στα ύψη. Θα αναλάβει τη διαβίωσή τους η Ευρώπη ή θα αναλάβει, θα αναλάβει να πείσει την Τουρκία την οποία χαϊδεύουν να δεχτεί την επαναπροώθηση στις χώρες από τις οποίες προέρχονται. Όσοι είναι πρόσφυγες και πληρούν τα κριτήρια του ΟΗΕ, βεβαίως η Ευρώπη να κάνει το καθήκον τους. Για τους υπόλοιπους πρέπει να επαναπροωθηθούν στις χώρες τους. Ευχαριστώ. <clears throat> Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, πριν δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο, διότι ορισμένα σημεία στην ημερήσια διάταξη και ορισμένες συζητήσεις απαιτούν από μένα τρομακτική αυτοσυγκράτηση. Θα ήθελα να υπογραμμίσω την έκκληση τη τελευταία της κυρίας Μωρέν Σάρτιε στο κλείσιμο της ομιλίας της και να συνοψίσω και πάλι. Εδώ πρόκειται για ανθρώπους. Μήπως το έχουμε ξεχάσει ε, ορισμένοι. Και ε, προσωπικά θεωρώ ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι παράνομος. Κανένας. δεύτερο, υπογραμμίζω ρητά ότι έχει μεγάλη σημασία να αποφύγουμε τον ανταγωνισμό μεταξύ των ανθρώπων. Να μην βάλουμε τους πρόσφυγες απέναντι στους πιο φτωχούς της κοινωνίας που ψάχνουν σπίτι ή χρειάζονται μια υποστήριξη. Άνθρωποι είναι όλοι και θα ήταν απάνθρωπο να τους ε, φέρουμε τον έναν αντιμέτωπο με τον άλλον. Τρίτον, θα πρέπει πραγματικά να προσέξουμε, να αφήσουμε ε, ξεχωριστά ε, την προσφυγιά από την τρομοκρατία, γιατί σε αυτή τη συζήτηση δεν συνέβη πάντα. Και για τα προσόντα και τις δεξιότητες θα ήθελα να παρακαλέσω την εισηγήτη να προσέξει πολύ προσωπικά ότι έχουμε ευρωπαϊκούς οργανισμούς που θα μπορούσαν να κάνουν πάρα πολλά για την αναγνώριση των προσόντων, για την προσέγγιση τους με τα ευρωπαϊκά για ανθρώπους που έρχονται εκτός Ευρώπης, αλλά έχουμε και επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια του κόσμου και έχουν ρυθμίσεις. Και εδώ ανήκει το υγειονομικό προσωπικό, γιατροί και ε, νοσηλεύτριες. Και θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει μια αντιστοίχηση και μια αναγνώριση των προσόντων τους. Και ένα τελευταίο, να σας στήσω να διαβάσετε ένα ανάγνωσμα. Η Financial Times και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό όταν εγώ αναφέρομαι στους Financial Times την Παρασκευή είχε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο άρθρο και συνέκρινε τον 30 κονταετή πόλεμο στη Γερμανία με τη σύραξη στη Συρία. Και είπα, όταν αυτό που είχε στην Ευρώπη το 17ο αιώνα και συντήρησε τον πόλεμο ήτανε η μόνιμη ανάμειξη των εξωτερικών μεγάλων δυνάμεων. Παρακαλώ προσοχή σε αυτό και να το λάβουμε υπόψη για να δούμε ποια διάσταση έχει η επιστροφή των προσφύγων. Αυτά ήταν μια ε, προσωπική παρατήρηση και σα ζητώ να με συμπαθάτε. Η Άννα Τομά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο, γιατί από χρόνο δεν πάμε παρακαλώ. Keine? Δεν έχετε σχόλια από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτό είναι ένα θέμα που είναι ευαίσθητο για μας και το συζητάμε με τη Γενική Διεύθυνση Home εσωτερικών υποθέσεων. Αυτό που μπορώ να πω τώρα από πλευρά Γενική Διεύθυνση Απασχόληση είναι ότι το εξετάζουμε, ότι σημειώνουμε τι παρατηρήσει των Ευρωβουλευτών, ιδιαίτερα όχι όσον αφορά την χρήση των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ήδη έχουμε αρχίσει να συζητάμε με τις χώρες μέλη πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν καλύτερα τα κονδύλια αυτά για να ενσωματώσουν στις κοινωνίες τους τους ανθρώπους αυτούς. Ε, αναφερθήκατε στις κατηγορίες. Πώς θα διαχωρίσουμε τους μετανάστες, τους πρόσφυγες, αυτούς που παίρνουν άσυλο μεταξύ τους. Πρέπει να στοχεύουμε καλύτερα τις δράσεις μας και τα κονδυλιά μας, πράγματι. Πάντω όχι μόνο η Γενική Διεύθυνση Απασχόληση, αλλά και άλλε υπηρεσίε Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζουν διαφορετικού τρόπου για να ενσωματωθούν καλύτεροι οι άνθρωποι αυτοί στι κοινωνίε μα και πώς θα συμπεριλαμβάνονται σε διάφορα προγράμματα, είτε ε, εκμάθηση γλώσσα, είτε επαγγελματική κατάρτισης κλπ. κλπ. Παίρνουμε πολύ στα σοβαρά το θέμα αυτό και βεβαίως και θα λάβουμε υπόψη μας τα αποτελέσματα των δικών σας εργασιών. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Για να δω λίγο τις προθεσμίες να σας πω. 15 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι για ε, τις τροπολογίες, τα είπε και η κυρία Μωρέν Σαντιέν. 18 Φεβρουαρίου θα ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή μας και στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ακόμα δεν έχουν ορίσει ημερομηνία. Ενώ στην Ολομέλεια θα πάει το Μάρτιο του 2016. Πάμε στο επόμενο θέμα, 10. Νέα εργαλεία εδαφική ανάπτυξη πολιτική συνοχή 2014-2020 Κουλυπού, το διαβάζετε. Η κυρία Σιόντροβα έχει το λόγο. Σόιντροβα. Thank you. Um, σας ευχαριστώ Πρόεδρε, να παρουσιάσω την έκθεση ε, για την οποία επί της ουσίας είναι υπεύθυνη Επιτροπή Ρέτζι για την ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση ITI στην τοπική ανάπτυξη των πρωτοβουλίων τοπικών κοινωνικών CLDD. CLLD μάλλον. Εδώ μας απασχολεί η διάσταση της απασχόλησης για αυτά τα εργαλεία χρηματοδότησης και θέλουμε να εντοπίσουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Πρώτα απ' όλα να τονίσω την δυνατότητα να έχουμε μία προσέγγιση bottom-up στην CLLD για την πρόθεση της εταιρικής ε, σχέσης, για τις κοινωνικές υποθέσεις και την απασχόληση. Εδώ έχουμε κληροδοτήσει το πρόγραμμα LEADER, ε, το προηγούμενο πρόγραμμα, που είναι πολύ σημαντικό για την απασχόληση στις τοπικές κοινότητες και την βιώσιμη ανάπτυξη υπαίθρου. Βλέπουμε ότι αυτά τα εργαλεία ε, σχετίζονται με όλα τα διευθυντικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε όλες τις περιοχές όπως οι αστικές. Βεβαίως, δυστυχώς, η πρωτοβουλία αυτής, η LLD, και η επένδυση ITI δεν έχουν την απαραίτητη προβολή και διαρθρώση με τις δυνατότητες χρηματοδότησης και οι αρχές που διαχειρίζονται τα εργαλεία αυτά δεν τα καθιστούν κατανοητά, επαρκώς κατανοητά στους ενδεχόμενους δικαιούχους. Εδώ θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κάτι μέλη να ασχοληθούν με το τι ενημέρωση χρειάζεται σε αυτό το τομέα. Η διάσταση της απασχόλησης και παρούσα είναι, αλλά θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω. Βάσει και τη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020, τα ευρωπαϊκά κονδύλια θα πρέπει την απασχόληση να την έχουν ω προτεραιότητα. Σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να επισημάνω την περιορισμένη χρήση των κονδυλίων από το Κοινωνικό Ταμείο, από το CLLD και το ITI. Έχω πολύ καλή συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών και τους δικούς τους εισηγητές για την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων όπου η συνεργασία μας βεβαίως και θα συνεχιστεί για να δούμε πώς αυτά τα δύο εργαλεία θα εφαρμοστούν καλύτερα στα κράτη-μέλη και θα παρακολουθήσουμε στενά μαζί με την Επιτροπή Ρέτζη την σωστή τους ε, εφαρμογή. Θα πρέπει να βρούμε τις σωστές παρατήσεις για την ενδιάμεση αναθεωρησή τους το 2017. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μας για την συνεργασία τους και την υποστήριξή τους και ε, αν για τα σχόλια ή τις τροπολογίες σας. Ευχαριστώ πολύ. Σκιώδης. 1,5 λεπτό έκαστος. Ο Γιώργη Πυρίνσκι πρώτος. Thank you, Chairman, and I would like to uh, express particular thanks. Ευχαριστώ να ευχαριστήσω εδώ την κυρία Σόντροβα για την ε, πολύ καλά διαδομένη γνωμοδότηση. Τρεις προτάσεις θα κάνω μόνον. Πρώτον, γνωρίζουμε ότι και το CLLD και το ITI είναι απολύτως αναγκαία για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Θα πρέπει να ε, ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κρατημέλη να προσφέρουν σε αυτές τις περιφερειακές αρχές ε, στήριξη για την υλοποίηση αυτών των πρωτοβουλειών. Δεύτερον, Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι και το ITI και το CLLD θα πετύχουν μόνον εφόσον αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις κοινωνικών υποθέσεων και απασχόλησης των συγκεκριμένων περιφερειών για κοινοθήτων. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό το να υπάρχει σωστή στοχοθεσία, στόχευση μάλλον, και τρίτον η περιορισμένη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για το CLLD και το ITI ήδη έχει προβλεφθεί, έχει καθοριστεί. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ότι θετικές για τα αστικά κέντρα, η οικοδόμηση θεσμικών δυνατοτήτων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είναι προτεραιότητες για να αντισταθμιστούν αυτές οι ελλείψεις. Ευχαριστώ κύριε Τρεμπέζιος. Α, ο κύριος Γκέρι και θέση Ευχαριστώ. Η κυρία Τρεμπέζιος ε, μου είπε να σας ευχαριστήσω κυρία Σόιδροβα, διαβάζω ένα κείμενο στα αγγλικά. Δεν έχω μεγάλες ανησυχίες ή προβλήματα με το περιεχόμενο της νομοδότησης. Συμφωνώ πολύ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτά που λέτε και το διοικητικό άχθος ε, και ε, τους μικρομεσαίους και τους ενεχομένους σε τοπικό επίπεδο. Θα ήθελα να τονίσω τα εξής η κοινοτική χρηματοδότηση δεν θα πρέπει να επιδοτεί εθνικές προσεγγίσεις, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιείται για επιπλέον ενίσχυση, συμπληρωματική και ενισχυτική των εθνικών προγραμμάτων, σύμφωνα με την απόφαση των κρατών μελών. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα θα πρέπει να προβλέπουν την απαραίτητη ευελιξία έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να εφαρμόζουν ε, τη δική τους ε, πολιτική ανάλογα με τις ανάγκες τους χωρίς να υπάρχουν υπερβολικοί έλεγχοι και λογιστικοί και άλλοι. Και οποιαδήποτε ε, αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ε, διαχείρισης των κονδυλίων στην απασχόληση και τα κοινωνικά δεν θα πρέπει να κοιτάει μόνο το κόστος και τον αριθμό των συμμετεχόντων αλλά και πώς αυτό έχει αντίκτυπο στην πραγματικότητα και μακροπρόθεσμα στη ζωή την εργασιακή και την ευρύτερη για να ε, έχει προτεραιότητες και να καταλαβαίνει με ποιο τρόπο πιάνουν τόπο αυτές οι προσπάθειες. Για την αναγνώριση λοιπόν και το σεβασμό των διαφέρων κοινωνικών και οικονομικών συστημάτων στα διάφορα κράτη-μέλη χρειάζονται προσπάθειες έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι η γραφειοκρατική διαδικασία δεν θα επιβαρύνει ιδιαίτερα τα κράτη-μέλη με άχρηστες και βαριές όσο και ακριβείς διαδικασίες. The focus from... Γιατί καμιά φορά αυτό μπορεί να αλλάξει την προσέγγιση και να φύγουμε από την προσέγγιση με βάση το αποτέλεσμα να κοιτάμε μόνο ε, τα κονδύλια. Ε, τέλος, για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, η ομάδα μας θα λέει ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί ε, μετά από αξιολόγηση αν χρειαστεί για να επαναχαραχθούν οι προτεραιότητες και η κατανομή των κονδυλίων σε διάφορες γραμμές του προπολογισμού σε σχέση με το, το TDP που εγκρίθηκε το 2014 θα πρέπει να παραμείνει η συνολική χρηματοδότηση όσο έχει χωρίς να αυξηθεί. Ευχαριστώ για την γνωμοδότηση αυτή και προσβλέπω στη συνεργασία με όλους τους σκιώδεις συγητές ε, και συντάκτες Σε ερχόμενες εβδομάδες. Ευχαριστώ λέει η κυρία Τρεμπέσιος. Ευχαριστώ. Ενάμιση λεπτό είπαμε. Το θυμίζω. Ο Ρίκε Καλβέσιος Σαμπον θα το καταφέρει σε είμαι βέβαιος. Ελπίζω, ναι. Πρόεδρε. Θα μιλήσω εκ μέρους της κυρίας Χάρκιν, που είναι η σκιώδης εισηγήτρια. Λέει λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για... Την εισηγήτρια μάλλον για το έργο της. Η κυρία Χάρκιν πιστεύει ότι η πολιτική συνοχής μπορεί να βοηθήσει όσον αφορά τις ευκαιρίες απασχόλησης. Και πιστεύει εκείνη, έτσι μιλάω στο όνομά της, πιστεύει ότι όταν η τοπική ανάπτυξη με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων χρησιμοποιείται ως εργαλείο, βελτιώνει την κατάσταση τοπικά και ανταποκρίνεται άμεσα στις τοπικές ανάγκες με τον καλύτερο τρόπο από ότι αν οι αποφάσεις λαμβάνονται κεντρικά. Όμως, ε, μία από τις πιο σημαντικές πτυχές όσον αφορά το CLLD και την ολοκληρωμένη δαφική επένδυση, ITI, είναι ότι πρέπει να υπάρχει βούληση από τις τοπικές αρχές και άλλους παράγοντες, ώστε η προσέγγιση είναι αυθεντική και οι τοπικές κοινότητες να μπορούν να αποφασίζουν μόνες τους για το τι είναι καλό και τι όχι. Συμφωνεί επίσης ότι η τοπική ανάπτυξη με την προβλήμα τοπικών κοινοτήτων είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη της υπαίθρου και μπορεί να βοηθήσει αντίστοιχα και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Προσβλέπει σε συνεργασία με την εισηγήτρια. Αυτά λέει η σκιώδης εισηγήτρια. Αλλά να προσθέσω και δύο προτάσεις εγώ. Μην ξεχνάμε ποτέ ότι η λύση είναι στη σωστή κινητικότητα. Μην πειράξετε την κινητικότητα. Πολύ καλά δίκτυα τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων είναι κάτι πολύ καλύτερο. Και θα επαναλάβω αυτό που είπε και ο Πρόεδρος, ότι είμαστε άνθρωποι. Δεν είμαστε δέντρα που γεννιούνται, ε, μεγαλώνουν και πεθαίνουν στο ίδιο μέρος. Παρατρίχα, περάσατε το 1,5 λεπτό. Ist Ουσιάζει η επόμενη ομιλήτρια, ωραία. Η Λαώρα Ατζέα. Παρακαλώ. Grazie Presidente. Με ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και για το σχέδιο γνωμοδότησης στην ε, συνάδελφο. Είναι πολλά τα σημεία αυτής της ε, γνωμοδότησης με τα οποία συμφωνούμε, όμως χρειάζονται κάποιες διευκρινήσεις. Εκεί όπου γίνεται λόγος για ανάπτυξη. Θα ήθελα να υπάρχει ε, ο όρος ανάπτυξη αλλά όχι απλώς οικονομική αύξηση, δηλαδή να υπάρχει και αυτή η ποιοτική διάσταση στην ενταφική χρήση των συγκεκριμένων αυτών εργαλείων. Πιστεύω ότι αυτή η βελτίωση θα είναι εύστοχη, διότι αυτό που θέλουμε είναι ανάπτυξη και βιώσιμη και συμμετοχική. Το να προβλέψουμε λοιπόν ένα τέτοιο όρο με ποιοτική χρειά είναι και πιο εύστοχο και πιο σκόπιμο. Πιστεύω ότι δεν είναι γνωστέ οι πρωτοβουλίε που υπάρχουν μέσω των εργαλείων αυτών σε, περιφερειακό επίπεδο. Θα έπρεπε λοιπόν κάποιοι να αναλάβουν την ενημέρωση, να είναι τα άμεσα σημεία επαφή ε, ω διαμεσολαβητέ μεταξύ Ευρώπη και εδαφικών των τοπικών και περιφερειακών φορέων. Θα έπρεπε λοιπόν να εκπαιδευτούν επαγγελματίε οι οποίοι να αναλάβουν αυτήν την ενημέρωση με την απαραίτητη κατάρτιση που είναι απολύτως αναγκαία. Πολύ συχνά έχουμε χρήση αναποτελεσματική των κονδυλίων σε περιφερειακό επίπεδο. Παρακολούθηση λοιπόν και τελευταίο σημείο να αναζητήσουμε να καταλάβουμε ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες στην πράξη, στις περιφέρειες και επαρχίες. Εκεί που γνωρίζουμε τι ακριβώς είναι απαραίτητο, το καταλαβαίνουμε να στοχεύσουμε καλύτερα και τη χρήση των συγκεκριμένων κονδυλίων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μωρά Σαχτσία έχει στήσει το λόγο. Και μετά η Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την συγκεκριά μας Μιγέλα Σουέντροβα για την έκθεσή της. Ήθελα να επανέλθω στο θέμα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και την μνήα που γίνεται για την ενδιάμεση αναθεώρηση. Αυτό σχετίζεται και με την παρατήρηση που έγινε προηγουμένως, αυτή που κάνατε και εσείς ο ίδιος, ε, κύριε Πρόεδρε, και που μας αφορά όλους, η ενδιάμεση αναθεώρηση δηλαδή. Θυμηθείτε ότι στην ε, συζήτηση για αυτή την περίοδο προγραμματισμού το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είχε αμφισβητηθεί Πολλοί ήταν οι συνάδελφοι που ήθελαν να συγχωνευτεί με τα ταμεία συνοχής χωρίς καμία διάκριση. Εδώ γνωρίζω πολύ καλά ότι μπορεί να υπάρξουν ανταγωνιστικές δράσεις, όμως θα πρέπει αντιφέτος να αξιοποιήσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο εδώ με αφορμή την έκθεση αυτή όπως και την προηγούμενη για να αποδείξουμε την χρησιμότητά του. Και τη στιγμή της ενδιάμεσης αναθεώρησης να το ε, ε, ενισχύσουμε. Πιστεύω ότι είναι ένας μοχλός, ένα εργαλείο μόχλευσης που θα πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ και να μην είμαστε αυτοί ως Ευρωπαϊκή Κοινωνικών, ε, Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων που θα κάνουμε πιο ευάλωτο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Μάλιστα. Προφανώς είναι αυτό και αυτονόητο. Τώρα, εξ Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάρτιν Ντεμπρέν. Good, um, good afternoon. Γεια σα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για τη γνωμοδότηση αυτή. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη και ενδιαφέρουσα για την εργασία μας. Θα ήθελα ε, εκ μέρου τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διευκρινίσω δύο πράγματα. Για την τοπική ανάπτυξη, 1,2 δις θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το επόμενο διάστημα. Αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα βρεθούν 1 δισεκατομμύριο για την περιοδευτή και από τα δύο ε, ταμεία λοιπόν ε, θα δοθεί ε, σημαντική ενίσχυση. Επίσης αναγνωρίζουμε ότι η κατάρτιση είναι πάρα πολύ σημαντική. Το έχουμε πει και στους ενδιαφερομένους και φτάνουμε σε δικαιούχους που για πρώτη φορά διαχειρίζονται κοινοτικά κονδύλια ευρωπαϊκά και δεν έχουν την απαραίτητη εμπειρία. Άρα χρειάζεται κατάρτιση και υποστήριξη για να μπορούν να τα διαχειρίζονται. Ένα λοιπόν από τα όσα κάνουμε, στείλουμε ένα δίκτυο αστικής ανάπτυξης παντού σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις ε, και με ε, ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις και υπάρχουν και άλλα δίκτυα για την τοπική αντίστοιχη ανάπτυξη. Αυτά μπορώ να σας πω εξ ονόμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ωραία. Σημειώνουμε λοιπόν 15 του στις 12 το μεσημέρι προθεσμία για τις τροπολογίες. 25 Ιανουαρίου ψηφίζουμε εμείς και η Περιφερειακή στις 15 του Φλεβάρι. Επόμενο θέμα, υπαριθμό 11, ισότητα των φύλων και ενδυνάμωση των γυναικών στην ψηφιακή εποχή. Η συγγήτρια είναι η Γιώτα Στάινροφ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η δουλειά μας ψηφιοποιείται και ο εργασιακός χώρος, το βλέπουμε αυτό και στην περιοχή μας και στην Επιτροπή μας. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό που δεν θα αλλάξει αν συνεχιστεί η κατάσταση είναι η ανισότητα, η ανισμεταχείριση ανδρών και γυναικών σε ό,τι αφορά τις καλά αμοιβόμενες θέσεις. Μιλώ για διακρίσεις βάρων των γυναικών. Ε, στα ηλεκτρονικά και στα ψηφιακά οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται και μάλιστα πολύ βαριά. Και γι' αυτό καλό τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασχοληθούν με ε, την υποστήριξη ε, στις εταιρείες των ψηφιακών επαγγελμάτων και των ζητημάτων της πληροφορική. Αυτό που θέλουμε περισσότερα κίνητρα να έχουν οι γυναίκες ε, ε, να ασχοληθούν με τέτοια επαγγέλματα, με ψηφιακά και ε, πληροφορική. Και να υπάρχει και σταδιοδρομία για να μπορεί να προσελκύει οι γυναίκες. Άρα χρειάζεται να εφαρμοστεί η οδηγία για ε, ε, μια ποσόστοση 40% υποχρεωτική ε, στα διοικητικά συμβούλια. Επίσης διαβίω εκπαίδευση, μετακπαίδευση, κατάρτιση, έτσι ώστε να προωθούνται και να προάγονται οι ψηφιακές δεξιότητες και να κλείσει ή να μειωθεί το χάσμα και το έλλειμμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα επικαλείται τις τόσες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν με την ψηφιοποίηση. Θέλει προσοχή εδώ τι είδους θέσεις εργασίες είναι αυτές και ποιες είναι αυτές. Να μην είναι τίποτα ε, δευτερεύουσες ε, πάρεργα, αλλά να μπορεί ο κόσμος να ζει από τη δουλειά αυτή. Οι γυναίκες επίσης θα πρέπει ε, να ε, μπορούν να συνδυάζουν τον επαγγελματικό με τον εργασιακό τους βίο και με άλλες μορφές εργασίας, τηλεεργασία κτλ. αλλά όχι με λιγότερη αμοιβή. Επίσης, ε, ε, θα πρέπει να υπάρχει προστασία των εργαζομένων και όχι μια ευελιξία κακώς νοούμενη που πληρώνουν τα σπασμένα οι γυναίκες. Ίσια αμοιβή λέμε πάντα για την ίδια εργασία για άνδρες και γυναίκες. Αυτό θα πρέπει να επικρατήσει και να ισχύει και στην ψηφιακή εποχή και επιτέλους να εφαρμόζεται. Επίσης, ε, προστασία της εργασίας και πάλι αλλαγές βλέπουμε στην ψηφιακή εποχή και μπορεί να είναι προς όφελος των γυναικών στη φροντίδα ε, των παιδιών τους. Υπάρχουν όμως τα θέματα του burnout, της κατάθλιψης και άλλα, όταν πρέπει να είσαι επί 24 ώρου βάσεως διαθέσιμος και ε, υπατμών για την υπηρεσία σου. Τα θέματα αυτά τα έχουμε ξαναδεί και στην προηγούμενη γνωμοδότηση και βρίσκουν τη συνέχεια τους ε, με τη σημερινή. Είναι ένα πρώτο πλαίσιο θα τα ξαναπούμε και σίγουρα θα μας απασχολήσει και πάλι αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κοσλόφσκα Ράγεβιτς. E, e, Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για την ε, έκθεση αυτή, η οποία περιλαμβάνει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Δεν θα αρχίσω από την ε, χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στις τεχνολογίες πληροφοριών. Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για έναν από τους τομείς όπου διαπιστώνουμε ότι υπάρχει διάκριση μεταξύ των δύο φύλων. Αυτό που εγώ βρίσκω πιο σημαντικό σε αυτήν την ε, έκθεση για την οποία εμείς κάνουμε γνωμοδότηση είναι η ψηφιοποίηση, η οποία τροποποιεί τα χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας στο σύνολό της, του περιβάλλοντος εργασίας και δημιουργεί νέες δυνατότητες, νέους τρόπους εργασίας, νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας. Όλα αυτά είναι μια πρόκληση για μας, για τη δικιά μας Επιτροπή. Οι νέες μορφές εργασίας έχουν πολλά θετικά, μπορούμε να φανταστούμε, γιατί σήμερα είναι πιο εύκολο, αν μη τι άλλο, να συνδυάσει κανείς την επαγγελματική με την προσωπική ζωή γιατί γίνεται πιο ελαστική η εργασία. Οπότε οι γυναίκες οι οποίες έχουν παιδιά και δυσκολεύονται να μπουν στην αγορά εργασίας ή άτομα ασθενή, ανάπηρα, χάρη στις νέες τεχνολογίες έχουν περισσότερες ευκαιρίες να συμμετέχουν στην αγορά αυτή εργασίας. Όμως όλα αυτά ελοχεύουν και κινδύνους. Και αυτά ακριβώ αναφέρει η γνωμοδότησή μας αλλά και η έκθεση. Διότι ο κίνδυνος είναι οι άντρες και οι γυναίκες που ασχολούνται με τις τεχνολογίες πληροφοριών είναι να βρίσκονται συνέχεια μπροστά στον υπολογιστή τους. Να μην απομακρύνονται ποτέ. Σε λίγο δεν θα είμαστε καν σε θέση να κλείσουμε όλα αυτά τα μηχανήματα που μας συνδέουν με το διαδίκτυο. Αυτό έχει να κάνει με τις νέες μορφές εργασίας. Κάποια πράγματα λοιπόν δεν διευκρινίζονται από πλευράς δικαίου. Υπάρχουν και κίνδυνοι όσον αφορά ε, το κοινωνικό δίκαιο, τον κώδικα δεδολογίας την εργασία κλπ. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας και σε κάτι άλλο. Γίνεται μια έκκληση εδώ για την διαβίου μάθηση οι ψηφιακές δεξιοτεχνίες δεν ε, ε, μαθαίνονται εξίσου εύκολα από τα άτομα κάποια ηλικία. Ο κίνδυνο λοιπόν για τα άτομα κάποια ηλικία που εξακολουθούν όμω να εργάζονται είναι να μην είναι σε θέση να ανταποκριθούν στι απαιτήσει τη ψηφιοποίηση και άρα σιγά σιγά να αποκλειστούν από την αγορά εργασία. Και αυτό έχει να κάνει κυρίω με τι γυναίκε γιατί αυτός ο ψηφιακός αναλφαβητισμός πλήττει περισσότερο τις γυναίκες. Γι' αυτό η διαβίου κατάρτιση έχει τεράστια σημασία ώστε να μπορούμε να χειριζόμαστε νέα μηχανήματα, νέα εργαλεία που χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες. Αυτές ήταν οι παρατηρήσεις μου, νομίζω, οι κύριες παρατηρήσεις μου τουλάχιστον. Στηρίζω πάντως την έκκληση αυτή που γίνεται, ώστε επιτέλους να γίνει πραγματικότητα η οδηγία αυτή για την ενδυνάμωση του ρόλου των γυναικών σε πιο ψηλά αξιώματα. Ευχαριστώ. Ο Τόμας Μάναρα προηγουμένως της να, να τελειώσουμε. Η Παλώμα Λόπες. Όλοι οι, υπόλοιποι, πολιτικέ υπόλοιπες πολιτικές ομάδες δεν μας έχουν δώσει ονόματα σκιωδών. Σηκώνει το κύριος Γκέρικε. Ναι, εντάξει, συγγνώμη. Παρακαλώ να πείτε στις πολιτικές ομάδες να δίναν κανένα ονοματάκι και να μας λένε εκ των προτέρων ποιος αντικαθιστά τους σκιώδεις ηγητές για να κανονίζουμε και το χρόνο, πώς θα το μοιράσουμε έτσι οργανωτικά. Εντάξει, ο κύριος Γκέρικε και η κυρία Ατζέα. Πολύ ωραία και μετά ο Τόμας Μαν. ή μήπως το γεγονός ότι δεν δίνουν ονόματα οι πολιτικές ομάδες είναι ότι η μήπω, το γεγονό οτι δεν δινουν ονοματα οι πολιτικέ ομαδες ειναι οτι φτάσει στην ομάδα μας, στην επιτροπή μας μάλλον. Η Οξφόρδη, το Πανεπιστήμιο, έκανε μια έρευνα για την Αμερικανική αγορά εργασίας και διαπίστωσε ότι στην επόμενη 20 ετία 47% των ε, εργασιακών σχέσεων ε, θα πληγούν. Στη Γερμανία 58% λέει αντίστοιχη μελέτη. Τα επόμενα χρόνια δηλαδή θα το βρούμε πάρα πολύ μπροστά μα και δεν είναι καθόλου επιπόλαιο το θέμα αυτό ή άσχετο και όχι μόνο δημιουργεί θέσει εργασία, αλλά θα έχει και πολύ μεγάλο κόστο. Ζητώ συγγνώμη για αυτή την παρένθεση Γκέρικε και Ατζέα. Στα αγγλικά διαβάζω την τοποθέτηση της και τη της μας. Ευχαριστώ την κυρία Στάιρουκ και να προτείνω και κάποια πράγματα. Θα ήθελε και όλη η να δει περισσότερα πρακτικά ζητήματα να ασχολούνται με τη βελτιοποίηση της ψηφιοποίηση των προσόντων για να ενδυναμωθεί και να ξεμπλοκαριστεί και η οδηγία για τη συμμετοχή γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Υποστηρίζουμε ε, όλους αυτούς τους ευγενείς σκοπούς, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε και τίποτα εθελοντικά μέτρα για να μπορούν οι γυναίκες να ανταποκρίνονται και στις ανάγκες της εκάστοτε πραγματικότητας σε εθνικό επίπεδο, αντί να ε, πιέσουμε να περάσει οδηγία. Θα χρειάζεται πολλή δουλειά στα κράτη-μέλη, έτσι ώστε τα μέτρα αυτά να πιάσουν τόπο και να ε, είναι υποφελή για τις γυναίκες. Η Σκιώδη Συγήτρια χαίρεται ε, για την αντίστοιχη δραστηριότητα που προβλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μια διοργάνωση της κυρίας Στάιρου. Και στην Επιτροπή Γυναικών η δική μας ε, εισηγήτρια θα είναι παρούσα εκεί για να συζητήσει αυτό το θέμα. Εμείς οι ε, συντηρητικοί και μεταρρυθμιστές πιστεύουμε ότι αν δημιουργηθεί ένα ε, περιβάλλον ευνοϊκό που θα ενισχύει τις επενδύσεις στην ψηφιακή επιθυμία θα είναι υπέρ των γυναικών με χαρά να βρούμε έναν τρόπο να εντάξουμε την τηλεεργασία και τις διάφορες ε, άλλες δυνατότητες για να μπορέσουν να εργάζονται περισσότεροι γυναίκες και άλλες ε, μειονεκτούσες ομάδες εργαζομένων. Θα κάνουμε και τροπολογίες αντίστοιχα στη γνωμοδότηση. Προσωπικά θέλω να προσθέσω στα γερμανικά ότι θα πρέπει να βάλουμε υπόψη εδώ τους γονείς, ιδιαίτερα τις μητέρες γιατί σε ό,τι αφορά την ψηφιακή αγορά και την ισότητα ε, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ε, ε, γυναίκες και για την ισότητα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τζέα. <coughs> Ευχαριστώ. Δεν έχουμε ορίσει σκιώδη γιατί και θα πρέπει να μιλήσουμε με τους συναδέλφους για να το επιλύσω. Θα υπάρξει συζήτηση πάντως για την έκθεση αυτή, γιατί είχαμε ασχοληθεί πάρα πολύ με την νέα ε, ψηφιακή αγορά. Το μόνο που θέλω να υπογραμμίσω εδώ, ε, σε αυτή την περίπτωση, και επιφυλασσόμενοι βεβαίω τη άποψη τη μελλοντική σκιώδη συγκεκριμένη είναι να δούμε τι θα γίνει ακριβώ με τι δεξιότητε. Η ψηφιοποίηση μπορεί να είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασία και για την επίτευξη ισότητα των φύλων. Όμω, εάν δεν εφαρμοστεί σωστά, εάν σωστά δεν δημιουργηθεί και ένα κατάλληλο πλαίσιο και πεδίο εντό του οποίου να μπορέσει να ενεργοποιηθεί, Υπάρχει κίνδυνος για μεγάλη μερίδα γυναικών που δεν θα έχουν απαραίτητες γνώσεις, ε, την απαραίτητη γνώση των ψηφιακών μέσων για να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις και τις νέες τεχνολογίες. Αυτέ είναι οι πρώτε αυτές είναι οι πρώτες μου ενθερμό Κατά πάσα πιθανότητα θα είμαι εγώ η σκιώδη εισηγήτρια, οπότε θα φροντίσουμε να υποβάλουμε τι παρατηρήσει μα μέσω των τροπολογιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Τόμα Μαν. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ Τόμας, αγαπητέ Πρόεδρε, έχεις δίκιο. Δεν είναι καθόλου επιπόλαιο το θέμα. Είναι πάρα πολύ κομβικό και κρίσιμο για το μέλλον. Καμιά φορά μου λείπει αυτή η θετική προσέγγιση. Είναι τεράστια ευκαιρία αυτό να μην λέμε μόνο άμυνα, αποκρούμε ε, τις προτάσεις, αντιδρούμε. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μια ισορροπία λογική. Δεν είναι όλα μαύρα. Υπάρχουν και φωτεινές πλευρές. Συμμετέχουν πολλές ε, επιτροπές ε, στην ψηφιοποίηση. Ο καθένας έχει τις δικές του αρμοδιότητες και η κάστοτε επιτροπή έχει τα χωράφια της. Είχα την ευκαιρία να συζητήσω ε, και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι 5-6 επίτροποι που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Εδώ, αγαπητή Γιούτα, ε, υποθέτω ότι θα κάνεις καλή έκθεση και ξέρω και με τους κοιόδης ηγητές θα συνεργαστείς πολύ καλά. Η μόνη παρατήρηση για τις γυναίκες γιατί είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό. Εγώ προέρχομαι από ένα τομέα που έχω άλλη εμπειρία. Ακριβώς οι γυναίκες που αξιοποιούν αυτή την ευκαιρία μπαίνουν πολύ πιο δυναμικά σε αυτούς τους τεχνολογικούς τομείς. Έχουν κατακτήσει τομείς ολόκληρους επαγγελματικούς. Και όχι μόνο είναι φάμιλες, είναι πολύ καλύτερες των ανδρών καμιά φορά. Άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οι γυναίκες είναι σε θέση να καλύπτουν αυτούς τους τομείς με δεξιότητες και προσόντα και δεν χωράει καμιά αμφιβολία αλλά να μην υπολείπονται και οικονομικά. Γι' αυτό έχουμε και εμείς αυτή την Επιτροπή εδώ απασχόλησης. Ε, θα καταλήξουμε σε κοινέ θέσει και ε, συμφωνώ. Λοιπόν, να λέμε ότι είναι και πολλές ευκαιρίες, όχι μόνο ε, δεινά, αλλά δεν είναι όλα αυτονόητα. Υπάρχουν και απειλές και προβλήματα αν δεν τα αντιμετωπίσουμε σωστά. Ως Επιτροπή Απασχόλησης λοιπόν, ανέκαθεν πατάμε και γερά στη γη και ξέρουμε τις πραγματικότητες. Ευχαριστώ. Προσβλέπω στην καλή συνεργασία και με τη Γιούτα Στάιν, που υποθέτω ότι σίγουρα είναι δεδομένη. Εγώ να δείτε, είμαι και εγώ πεπισμένος. Παρακαλώ να μην με παρεξηγήσετε. Δεν είναι τίποτα να αποκρούσουμε ή να αποδεχθούμε. Αυτό είναι γεγονός. Θα το βρούμε μπροστά μας. Δεν υπάρχει απόκρουση. Ε, και παντού και στην παραγωγή και στα γραφεία εμείς θα πρέπει να δούμε πώ θα το ε, αντιμετωπίσουμε, όχι πώς θα το αποκρούσουμε, δεν μπορούμε να το αποτρέψουμε. Πώς θα δημιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις για να δουλεύει ο κόσμος. Η κυρία Μωράν Σαρτιέ. Euh, Ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω την κυρία Στάιρουκ. Θα ήθελα στην παρέμβασή μου να ακολουθήσω την κατεύθυνση με την παρατήρησή σας. Θέλουμε αυτή η πλήρης συμπερίληψη των νέων τεχνολογιών στον επαγγελματικό βίο να γίνει σωστά. Από την οπτική γωνία της ισότητας των ε, φύλων, ανδρών και γυναικών, υπάρχουν δύο σημεία στα οποία θέλω να σταθώ και θα προτείνω σχετικά τροπολογίες. Από τη μια, η ισότητα των επαγγελματικών ευκαιριών και σταδιοδρομιών μεταξύ ανδρών και γυναικών, διότι υπάρχουν νέοι κλάδοι που αναπτύσσονται και ήδη υπάρχουν ανισότητες στους παραδοσιακούς τομείς τους. Νέους τομείς θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ε, αποφασισμένοι για να υπάρχει ισότητα στι επαγγελματικέ ευκαιρίε ανδρών και γυναικών. το δεύτερο σημείο στο οποίο θέλουμε να εμείνουμε είναι οι νέε μορφέ εργασία. Αυτέ οι νέε μορφέ εργασία σημαίνουν ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το πώ θα συνδυάζονται ο επαγγελματικό και ο οικογενειακό βίο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε τίποτα. Uh, το όνομά σας παρακαλώ. Um, Ευχαριστώ Πρόεδρε, απλώ να σα πω ότι παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή τι συζητήσει και το θέμα αυτό το ε, λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Όπω αναφέρατε και όπω ανέφερε και ένα ε, βουλευτή μα για την ε, στρατηγική τη ε, νέα ψηφιακή αγορά, δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή στο να υπάρξει ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά και για τους ανθρώπους με αναπηρία που θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις ψηφιακές ευκαιρίες. Υπάρχουν νέες μορφές ε, εργασίας όντως που προέρχονται λόγω της... προκλήθηκαν από την ψηφιακή επανάσταση. Θα έρθει στιγμή να τα συζητήσουμε όλα αυτά και θα μελετήσουμε πολύ προσεκτικά το θέμα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Άλλαξε κάτι με τις ε, προθεσμίες. Για την κατάσταση τροπολογιών δεν είναι 9 Δεκεμβρίου, αλλά 10 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι λήξη προθεσμίας, 10. Ε, ε, Εμείς θα ψηφίσουμε 25 Ιανουαρίου και στην Επιτροπή Γυναικών 17 Φεβρουαρίου. Στην Ολομέλεια είδομεν. Δεν είναι ακόμα ορισμένος. Λοιπόν, επόμενο θέμα, στη μέση διατάξη 12 επίτευξη του στόχου κατά της στόχες δεδομένων των αυξανωμένων εξόδων των νοικοκυριών. Ο Τάμας Μέζεριτς έχει το λόγο, εισηγητής μας. Τάμας, αν γίνεται 7 λεπτά σου φτάνουν, συνολικά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Όντως θα προσπαθήσω να ολοκληρώσω έγκαιρα. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ τους κοιόδης εισηγητές και όλους τους συναδέρφους για τις τροπολογίες που έχουν υποβάλει, πολύ άριθμες. Θα αναφερθώ σε κάποιες από αυτές, αλλά όχι βέβαια σε όλες, γιατί είναι πάρα πολλές συνολικά. Θα αφήσω και τους κοιόδης εισηγητές να αναφερθούν σε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τις τροπολογίες και πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε ετοιμάσει συμβαστικές τροπολογίες και στις συναντήσεις που θα έχουμε με τους χειόδους συζητητές θα συζητήσουμε πάνω σε αυτές. Υπάρχουν τώρα διάφορες τροπολογίες οι οποίες ε, μεγαλώνουν το κείμενο, το προεκτείνουν προς διάφορες κατευθύνσεις. Θυμόσαστε την πρώτη φορά που συζητήσαμε εδώ Είχα πει ότι είναι όλες ευπρόσδεκτες, γιατί έτσι καλώς το σχέδιο έπρεπε να είναι περιορισμένο όσον αφορά την εκτασή του και δεν μπορούσαμε να τα συμπεριλάβουμε όλα. Οπότε καλό αυτό. Με τις περισσότερες συμφωνώ. Με κάποιες άλλες προεκτάσεις νομίζω ότι δημιουργούν κάποια προβληματάκια στο κείμενο, αλλά θα ξεπεραστούν. Είμαστε στην ίδια γραμμή όταν μιλάμε για την φτώχεια και για τα αυξανόμενα έξοδα των οικοκυριών, που είναι ένα περίπλοκο ζήτημα. Δεν πρέπει να το περιορίσουμε απλουστικά. Όχι. Πρέπει να δούμε τις διάφορες πτυχές χωριστά, σε χωριστά κείμενα, σε χωριστές παραγράφους το καθένα. Εμείς οι πράσινοι επίσης Είμαστε απολύτως υπέρ της αρχής της επικουρικότητας. Πιστεύουμε ότι τα θέματα στα οποία τοπικά λύνονται καλύτερα πρέπει να λύνονται τοπικά. Και ότι σε ένα άλλο επίπεδο, σε ένα άλλο επίπεδο. Γι' αυτό προς αυτή την κατεύθυνση θα εξετάσουμε και όλες τις τροπολογίες, αν συνάδουν με αυτή την αρχή. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε παντού σε συμβασμούς. Υπάρχουν πολλές διάφορες νέες ιδέες πάντως από τους σκιώδεις. Δεν μπορώ τώρα να σας παρουσιάσω ένα πλήρη κατάλογο. Όμως θέλω να αναφερθώ στην κοινωνική κατοικία. Είναι ένα από τα ζητήματα που συμπεριλαμβάνουμε με όλες τις, τις το κατά πόσο υπάρχουν διαθέσιμα τέτοια σπίτια, κοινωνική κατοικία δηλαδή παντού, και οι κρατικές υπηρεσίες έχουν ένα ρόλο κλειδί να παίξουν. Επίσης, το θέμα των άστεγων. Και αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Παρόλο που καθαρά τεχνικά και απόλυτα μπορεί να φαίνεται να είναι εκτός του εύρους της έκθεσης αυτής, όμως είναι συνδεδεμένο γιατί τα νοικοκυριά που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας καταλήγουν άστεγα. Και αυτό σημαίνει σε πολλές χώρες μέλη. Τέλος, θέλω να προσέξουμε όλοι το εξή. Κάποιες από τις τροπολογίες χρειάζονται διαφορετική διατύπωση για να συμπεριληφθούν στο κείμενο. Οπότε θα ήθελα να σας την υπομονή σας για να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε το κείμενο κατάλληλο ώστε να συμπεριληφθούν και οι τροπολογίες αυτές. Επαναλαμβάνω πάντως ότι ευχαριστώ όλους τους σκιώδες και όλους τους συναδέρφους για τη βοήθειά τους για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Το έχω ξανακούσει αυτό με τις αναδιατυπώσεις των κειμένων. Μου φαίνεται γνωστό. Μια παράκληση πρέπει να φύγει η Λάουρα Ατζέα. Κανονικά θα να πάρει τρίτη το λόγο. Θα παρακαλώ τους συναδέλφους Άρνε Γκέρικε και τον ε, Κλοντ ε, Γολέν αν αφήνουν να πάρει το λόγο η Λάουρα πρώτη. Ναι. Η Λάουρα. Σας Ευχαριστώ για την ευγένεια, αλλά όπως και συνάδελφος, ε, ο συνάδελφος Γερή, είμαι στην αντιπροσωπεία για τις χώρες ΑΚΕ και πρέπει να φύγω γρήγορα. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Μεσρίτ Ταμάς για την ε, ε, διάθεσή του να έχουμε ένα τέτοιο κείμενο αποφασιστικό, διότι υπάρχουν πολλά σημεία που χρήζουν δυναμική τοποθέτηση από τη δική μα Επιτροπή. Έχουμε ήδη ετοιμάσει τροπολογίε βάσει των ενδείξεων που είχαμε δώσει σε προηγούμενη συζήτηση. Σε κάποιε πτυχέ καταλαβαίνουμε ότι μπόρεσε να ε, μεγαλώσει το πεδίο δράση μα, αλλά θα πρέπει να δούμε και τι συμβαστικές προτάσεις θα βρεθούν. Οι πρώτες ιδέες που μας υποβλήθηκαν ελπίζουμε ότι θα μας επιτρέψουν να οδηγηθούμε σε σημείο συμφωνίας. Η μείωση του κόστου των δαπανών για την ενέργεια είναι μια ε, σημαντική πτυχή. Αυτό το έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, απόλυτη ανάγκη να προβλέψουμε και στέγη για τους ε, αστέγους. Ξέρουμε ότι σήμερα ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, οι άστεγοι, είναι μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, αλλά Υπάρχουν και άλλα επιχειρήματα που προβάλαμε, όπως η ανάγκη του ελάχιστου προστατευμένου μισθού, εισοδήματο εισοδήματος και βεβαίως θα φροντίσουμε με τις συμβαστικές προτάσεις να επεξεργαστούμε μια κοινή θέση. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους. So, Ευχαριστώ πολύ κύριε Euh, euh, Ευχαριστώ. Πολλές συντροπολογίες. Ευχαριστώ τον εισηγητή για τη δουλειά που έχει κάνει μέχρι τώρα αλλά και για τη δουλειά που θα χρειαστεί να κάνει ακόμα για τις τροπολογίες αυτές. Πάντως εμείς θα βοηθήσουμε ώστε να καταλήξουμε σε μια έκθεση η οποία να είναι συνενετική και όσο γίνεται πιο πυκνή. Από πλευρά του ΕΛΚ όντως υποβάλαμε διάφορες τροπολογίες δεν θέλω να τις αναφέρω εδώ, θα μας έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο, θα τις συζητήσουμε με τον εισηγητή και τους άλλους σκιώδεις. Πάντως ένα από τα βασικά στοιχεία της συζήτησης είναι πού πρέπει να βρίσκεται το κατάλληλο επίπεδο απόφασης και ποιες είναι οι καταλληλότερες πολιτικές. Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ένα εργαλείο δεν μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό το οποίο επιθυμούμε Επίσης, χαίρομαι που διευρύναμε το εύρος, που αναφερθήκαμε και στην ενέργεια και που μπορέσαμε να ασχοληθούμε και με το θέμα της επικοινωνίας και των τεχνολογιών ε, πληροφορικής. Θέλουμε να καταλήξουμε σε μια έκθεση όσο γίνεται πιο συνετικά, όχι ως αυτό σκοπό, αλλά γιατί αυτό χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε μια στήριξη όσο γίνεται περισσότερο ευρεία και στην Επιτροπή μας εδώ, αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οπότε διαβεβαιώνω τον εισηγητή ότι θα έχει τη στήριξή μας. Ευχαριστώ πολύ. Α, τώρα βρήκαμε και εισηγητέ. Γιούταν Στάιροκ, ε, αντικαθιστά του Ισοσιαλίστε. Ναι, δυστυχώς ε, κολλείται η δική μας και όλη η εισηγήτρια και ε, με παρακάλεσε η κυρία Μία Πέτρα Κομπούλα να, να ευχαριστήσουμε. Ε, θέλουμε όλοι οι άνθρωποι να έχουν ελάχιστο εισόδημα ε, και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για να αποτραπεί ο κοινωνικός αποκλεισμός και η ένδια. Το λέμε και στις τροπολογίες μας. Αλλά Δεν θα πρέπει να κοιτάμε μόνο τους ανέργους. Υπάρχουν και εργαζόμενοι φτωχοί. Δυστυχώς με ραγδαία ε, αύξηση αυτό το φαινόμενο. Δεν είναι μόνο οι άνεργοι, οι φοιτητέ, οι ηλικιωμένοι, οι μονογονιακές οικογένειες, άρρωστοι. Πάνω από 50 εκατομμύρια είναι οι άνθρωποι στην Ευρώπη που ζουν σε συνθήκες ενεργειακής στόχιας. Είναι το 30% όλων των οικοκυριών και εμείς θέλουμε σε τοπικό, περιφερειακό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να περιοριστεί και να εξαλειφθεί τελείως η ενεργειακή φτώχεια. Γι' αυτό χρειάζονται μέτρα ενεργειακής απόδοσης και για το λιανικό εμπόριο, αλλά για όλα αυτά χρειάζεται ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την καταπολέμηση ε, αυτής της ενεργειακής στόχιας. Δεν θα πρέπει να είναι πανάκριβα τα τιμολόγια του νερού ε, ή ε, του ηλεκτρικού ή της θέρμασης. Δηλαδή δεν πρέπει ο κόσμος να ε, πρέπει να επιλέγει ανάμεσα σε ένα ζεστό σπίτι ή σε ένα ζεστό πιάτο φαΐ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και για μας και για τον εισηγητή και για άλλους είναι πολύ σημαντικό και το ζήτημα της κοινωνικής κατοικίας φυσικά και δεν θα πρέπει ποτέ να πέσει στο βωμό της λιτότητας μια αποτελεσματική κοινωνική πολιτική είναι το σημαντικότερο ε, εργαλείο για να αποτραπεί η ενεργειακή φτώχεια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αρνέ Γκέρικε. Τελευταία φορά πρόεδρε για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ και ήταν εισηγητή. Αν δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη και ποιο ε, είναι το προστιθέμενο όφελος για τους πολίτες, εντάξει, αλλά δεν είναι μόνο προς όφελος των επιχειρήσεων. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι να βοηθήσουμε τις οικογένειες και η άχρηστη ευρωπαϊκή γραφειοκρατία επιβαρύνουν την τσέπη και τον οικογενειακό προπολογισμό των πολιτών μας. Θα πρέπει να έρθει η γραφειοκρατία και τονίζω, η φτώχεια στις οικογένειες δεν προκύπτει μόνο από τα πολλά έξοδα. Στη χώρα μου τα παιδιά για πολύ κόσμο ε, είναι κίνδυνος να πέσουν στη φτώχεια. Όποιος σήμερα ε, στο σπίτι του ανατρέφει τρία και τέσσερα παιδιά ε, κάνει πολύ περισσότερα για να αναπτυχθεί η κοινωνία και δίνει και εισφορές. Ε, στις περισσότερες χώρες όμως δεν προβλέπεται τίποτα για όσους ανατρέφουν τα παιδιά τους στο σπίτι. Εδώ και 30 χρόνια το δικό μου κόμμα θέλει να δοθεί ε, μισθός ε, στη μητέρα ή στο γονέα που μεγαλώνει τα παιδιά του. Μισθός, ανατροφής, όχι επίδομα, όχι φιλοδόρημα. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν για το μέλλον της κοινωνίας. Και να είναι κοινωνικό αυτό όπως και η σύνταξη. Μισθός λοιπόν ανατροφής και όχι επιδόματα. Ε, θα κάνουμε τις τροπολογίες μας και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τους συζητητές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ο Ενρίκε por Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για την δουλειά που αρχίζει με τόσε πολλέ τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Θα δουλέψουμε κι εμείς πάνω στις συμβαστικέ προτάσεις. Οι ιδέε τη ομάδα μου, της ΣΑΛΤΕ, είναι στην γραμμή της διεύρυνσης του ορισμού του ότι είναι φτώχεια. Φτώχεια είναι κάτι που αντιμετωπίζεται με τις κοινωνικές πολιτικές η ανεργία από τις οικονομικές πολιτικές. Η φτώχεια είναι εδώ και τώρα. Δεν πρόκειται για μια δομή. Με κοινωνικές πολιτικές αντιμετωπίζεται. Η φτώχεια είναι και ενεργειακή βέβαια, αξίζει τον κόπο. Αλλά έχει και άλλους παράγοντες η φτώχεια που την επηρεάζουν. Το να μπορεί να έχει κανείς ένα σπίτι και να μην είναι άστεγος ή να μπορεί να στέλνει τα παιδιά του στο σχολείο. Η καταπολέμηση της φτώχειας ε, λοιπόν είναι αυτό που μας απασχολεί. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε και ένα ελάχιστο εισόδημα που να προσαρμόζεται στην κατάσταση της κάθε χώρας. Εγώ έχω μιλήσει με πολλούς τέτοιους ανθρώπους που βρίσκονται στην φτώχεια και τελικά δεν μπορούμε να λέμε των παιδιών, ενεργειακή, δεν ξέρω εγώ τι. Φτώχεια είναι, μία είναι η φτώχεια. Και οι άνθρωποι θα μπορούν να, είναι, να ζουν αξιοπρεπώς αν έχουν ένα ελάχιστο εισόδημα. Αυτή λοιπόν είναι ενδιαφέρουσα ιδέα για το ελάχιστο εισόδημα. Και άλλες ιδέες είναι ενδιαφέρουσε. Αλλά πάντα έχοντας υπόψη μας το ότι η φτώχεια δεν είναι μόνο θέμα τεχνικό, προστασία από την ενεργειακή ένδυα κτλ. Είναι γενικότερο και εξαρτάται από το κατά πόσο υπάρχει ένα ελάχιστο εισόδημα για το κάθε νοικοκυριό. Αυτό λοιπόν και άλλα πράγματα που χειρίζεται πολύ καλά ο εισηγητής μας βρίσκουν ε, σύμφωνο. Σίγουρα θα καταλήξουμε σε ενδιαφέρουσες συμβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα έχω μόνο τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος ε, Κριστόφ Μαρσάλ Ντομπρά. Σύντομα, αν επιθυμείτε, δεν είναι υποχρεωτικό. Επιθυμείτε. Yes. Lepo. Yes, hello. Yeah. Uh, yes, so, uh, well, the commission thanks. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευχαριστεί όλους τους μετέχοντες. Ιδιαίτερα όσοι έχουν ασχοληθεί με τις ε, πρωτοβουλίες κοινωνικής ένταξης και με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση. Προκειμένου να ολοκληρώσουμε την Νομισματική και Οικονομική Ένωση, πρέπει να προβλέψουμε για ένα πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην κοινωνική δικαιοσύνη και τα προγράμματα κοινωνικής ε, ε, ένταξης. Ευχαριστώ πολύ από τις συντομότερες τοποθετήσεις στην Επιτροπή μας αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πριν φύγετε όλοι, θα ήθελα να σας πω το εξής. 6.30 ώρα έχουμε ένα κοκτέιλ εδώ στον τρίτο όροφο του παρόντος κτηρίου ε, για να γιορτάσουμε το τέλος της ε, χρονιάς. Όσοι μπορείτε να συμμετάσχετε, όλοι οι υπόλοιποι που δεν είστε συντονιστές, παρακαλείστε να αποχωρήσετε το συντομότερο για να αρχή συνεδριάς των συντονιστών. Η γραμματεία μου έχει ετοιμάσει ημερήσια διάταξη για τους συντονιστές για δύο συνεδριάσεις. Όπως ε, όταν έκανα άλμα εις ύψος και μου βάζω προπονητής όλο και πιο ψηλά τον πύχη να πηδήξω. Λοιπόν, να δω πώς θα τα προλάβουμε. Παρακαλώ να ε, περάσουμε γρήγορα στη συνεδρίαση των συντονιστών για να προκάνουμε και όσους δεν σας ξαναδώ, καλές γιορτές. Και όπως λέμε στη Γερμανία να σας πει καλά το νέο έτος. Ε, και να περάσετε πολύ ωραία, να ξεκουραστείτε και θα τα ξαναπούμε στις 11 Ιανουαρίου ε, από τις 3 μέχρι τις 6.30.